Καλημέρα σας, να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας με την έκθεση της συναδέλφου Νίπλερ για την περιαγωγή, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τη συνεδρίαση των συντονιστών Εχθές το πρωί έγινε η συνεδρίαση των συντονιστών και οι αποφασίσεις που ελήφθησαν είναι οι εξής. Οι κύριοι Μάρτιν Όαρ και Τάμιστ ορίζονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΣΕΡ. Τα μέλη που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, καλούνται ε, για να αναφέρουν στην Επιτροπή Ήτρε ε, δύο φορές το χρόνο. Επιβεβαιώθηκε επίση η αντιπροσωπεία στη Βραζιλία και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να μας υποδείξουν τους συμμετέχοντες μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και το ταξίδι θα γίνει Ε, την ε, Δευτέρα 2 Απριλίου όταν θα ξεκινήσουν και οι εργασίες. Ε, η Γραμματεία θα επαληθεύσει τις προτάσεις που θα γίνουν με βάση τα κριτήρια που συμφωνήσαμε. Οι συντονιστές επίσης επιβεβαίωσαν την απόφαση που ελήφθη στην αρχή της θητείας για τον ορισμό των εκπροσώπων της Επιτροπής Ήτρες στη ΣΤΟΑ. Οι συνάδελφοι Ρούμπικ, Μαντορέλ, ε, Γιάνσεν και το Ζασκόφσκι είναι τα μέλη της ΣΤΟΑ. Και επίσης για τις ακροάσεις, ε, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει ακρόαση για το ορίζον 2020 στις 20 Μαρτίου του 2012 και για το πρώτο εξάμεινο του 2012 η Επιτροπή μας θα οργανώσει τρεις ακροάσεις, μία για το ορίζον 2020, μία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μία για την ψηφιακή ατζέντα. Κατόπιν, στο δεύτερο εξάμεινο υπάρχει δυνατότητα να διοργανωθούν και κάποιες άλλες ακροάσεις για την πολιτική του διαστήματος, για τις ευφυείς πόλεις ε, και τις ε, καινοτόμες τεχνολογίες. Όσον αφορά τώρα τις μελέτες και τα εργαστήρια, καλούνται όλες οι πολιτικές ομάδες να αποστείλουν στη Γραμματεία μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου προτάσεις. Στη διάρκεια της συνεδρίασης μοιράστηκαν και τέσσερις εκθέσεις. Το πρόγραμμα Horizon 2020 στο ΕΛΚ, το πρόγραμμα για την έρευνα της Ευρατόμ στους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ινευρέπη των Συντηρητικών και Δημοκρατών και η πυρηνική ασφάλεια στους φιλελευθέρους. Όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις, θα οριστικοποιηθούν μετά από τη διαβούλευση μεταξύ των συντονιστών. Αυτά λοιπόν ενημερωτικά από πλευρά μου για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες ε, της σημερινής ημέρας βάσει της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης προβλέπει τη συζήτηση για την έκθεση της συναδέλφου Νίμπλερ για την ε, περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης. Παρακαλώ κύριε Νίμπλερ. Συγγνώμη. Μετά θα λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώ αμέσως και ασχολούμαι με το πρώτο θέμα. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η ισχύουσα κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες για την έκθεσή μου 359 τροπολογίες στο σύνολό τους οι οποίες έχουν διατυπωθεί μέχρι στιγμής και προσπάθησα στη συνέχεια με τη βοήθεια της γραμματείας να προβώ σε ε, συμβιβαστικές τροπολογίες κατά τρόπον ώστε να απλοποιήσω το θέμα γιατί όλες ε, οι τροπολογίες συγκεντρώνονται σε τέσσερα βασικά ε, σε τέσσερα τέσσερις βασικές ε, θεματικές ενότητες τις οποίες θα αναφέρω τώρα ε, και θα μου πείτε αν κάπου δεν κατάλαβα ε, ε, ε, την, ιδέα σωστά. Οι ιδέες έχουν ήδη διανεμηθεί από το Κοινοβούλιο και φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι έχουν όλοι λάβει τις συμβιβαστικές τροπολογίες μου. Οι αλλαγές οι οποίες δεν υπάρχουν στις τροπολογίες νομίζω μπορούν να λευκανθούν μέσω της τροπολογίας και έτσι θα περιοριστώ στις 15 συμβιβαστικές τροπολογίες ε, έχοντας ρίξει και ένα μάτι προς το Συμβούλιο γιατί προσπάθησα ε, να καταλήξω σε ε, μία ε, ε, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι στη συνέχεια θα μπορέσει ο νέος ο κανονισμός να ισχύσει γιατί είναι πλέον ώρα να μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε και γι' αυτό θα προτείνω να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Πρόκειται για το ε, θέμα του roaming, της περιαγωγής. Ε, καταρχήν όσον αφορά τα ανώτερα επίπεδα τιμής χοντρικής και λιανικής όπου έχουν ε, διατυπωθεί διάφορες προτάσεις και ορισμένοι ζητούν ακόμη πιο αυστηρές ε, ιδέες από ότι εγώ ε, έχω <clears throat> προτείνει και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν συμφωνήσει με την δικιά μου πρόταση. Θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα να βρω μία μέση τιμή και ελπίζω ότι κατόπιν αυτού θα έχω αποκλίνει τις τιμές διότι ε, για να το επιτύχω αύξησα λίγο τις τιμές ε, για τα SMS κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να μείνουμε σε έναν μέσο όρος και ε, η πρόταση αυτή προσπαθεί να λάβει υπόψη όλες τις προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί. Κατέληξα λοιπόν σε αυτή τη μέση τιμή και θα μου πείτε εάν είναι εύστοχη η λύση που προτείνω ή όχι. Όσον αφορά την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς που συναποφασίζει στον τομέα αυτό και αυτή <coughs> θα χρειαστεί να εκφράσει τη γνώμη τους και αύριο θα ψηφιστεί εκεί η γνωμοδότηση και οι τιμές είναι υψηλότερες από αυτές τις οποίες έχουμε προτείνει εμείς. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ μιλάμε για ανώτατες τιμές θα πρέπει <clears throat> να καταλήξουμε σε μία λογική μέση λύση κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να πάμε στις ε, συνδιαλλαγή με μια ισχυρή πλειοψηφία και εδώ αναφέρομαι εις ε, τις τροπολογίες 19, 11, 12, 13 και 14. Ε, θα επανέλθω λοιπόν ε, στο θέμα αυτό όταν θα έχω προτάσεις σας. Ο δεύτερος τομέας που με απασχόλησε ήταν τα διαρθρωτικά μέσα και εδώ διαπιστώνω ότι τα προτινόμενα μέτρα αυτά στηρίζονται από πολλούς και εκεί συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι είπαν ότι θα έχουν, θέλουν πολύ χαμηλό ανώτατο πλαφόν ε, και άρα να μην υπάρξουν διαρθρωτικά μέτρα αλλά ε, υπάρχει και ε, ένα μέρος των Ευρωβουλευτών που συμφωνεί με αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα και επίσης υπάρχει και ένα θέμα άλλο το οποίο τίθεται το roaming profile δηλαδή τα τεχνικά μέτρα και μία ε, έκδοση της εφαρμογής αυτών των διατάξεων ε, έχουν ε, επίσης επικροτηθεί και προτείνεται να ληφθούν τα δύο διαρθρωτικά μέτρα και γι' αυτό έχω καταλήξει σε μία συμβιβαστική τροπολογία τέσσερα επί του θέματος. Η άλλη ιδέα ήταν να υπάρξει ένα local breakout στην έκθεση. Δηλαδή υπάρχουν επί του θέματος αυτό πολλές τροπολογίες από συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες και σκέφτομαι ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ λογική, δηλαδή καταρχήν να συμφωνήσουμε με τα δύο μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια να δεχθούμε και το local breakout και τώρα έχω διατυπώσει την, ε, την συμβιβαστική τροπολογία 6 που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το συγκεκριμένο θέμα και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω ε, αγαπητοί συνάδελφοι είναι η συμβιβαστική μου πρόταση 5 ε, ε, σχετικά με το opt-out και την σχετική ρήτρα όπου έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις δηλαδή αν ένας πάροχος δεν υποχρεούται να προβεί σε διαρθρωτικά καμετρα μετρα μέτρα, δηλαδή μέτρα opt-out, εάν οι τιμές, του, ε, ε, οι τιμές που προσφέρει για τις επικοινωνίες στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό είναι συγκρίσιμες και πολύ κοντινές. Δηλαδή όταν το εθνικό τιμολόγιο με το τιμολόγιο του roaming είναι πολύ κοντά δεν χρειάζεται το opt-out και ε, θεώρησε ότι η ιδέα αυτή ε, είναι περίεργη διότι εμείς θέλουμε μία ε, ελεύθερη αγορά να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ ε, της, των τιμών εσωτερικού και εξωτερικού και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε ε, σε μία διεύρυνση της αγοράς η οποία πρέπει να ανοίξει και πιστεύω ότι με την λύση αυτή δεν επιτυχάνεται γι' αυτό και πρέπει να το ξανασκεφτούμε ε, θα αναμείνω οι συνάδελφοι να μου δώσουν και άλλες ιδέες εάν θέλουν αλλά γενικώ Θέλω να ευχαριστήσω για τις πολυάριθμες τροπολογίες που υποβλήθησαν, εκ των οποίων πολλές βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και ελπίζω ότι τώρα στη συζήτηση θα, υπάρξει, ε, θα υπάρξουν προτάσεις για συμβιβαστικές ιδέες κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε σύντομα να ψηφίσουμε και να προχωρήσουμε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Νίπλη. Ξέρετε ότι στις 10 θα ψηφίσουμε, επομένως ε, ε, θα μιλήσουμε μέχρι τις 10, γι' αυτό ε, εάν χρειαστεί θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε μετά από την ψηφοφορία. Μία ενημέρωση τώρα από τη Γραμματεία όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τις μοιράσουν, διότι εχθές τελείωσε η συνεδρίαση, επομένως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να διανύμουν τα συμβαστικά κείμενα. Αυτό ήθελα να σας πω ενημερωτικά. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Έχουμε τους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Γκέμπελς θέλει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι λυπάμαι που ο πολύ αποτελεσματικός μας πρώην πρόεδρος Ρόιλ δεν είναι πια πρόεδρος επιτροπής μας. Ε, ε, σας συγχαίρω για την εκλογή σας και είμαι βέβαιος ότι οι εργασίες μας ε, θα συνεχίσουν εξίσου ομαλά. Θα ήθελα καταρχάς την καλή μου φίλη Αγγέλη Κανίμπλερ να την ευχαριστήσω για όλη την καλή της δουλειά χθες το βράδυ. Ε, είχαμε μία συνάντηση μαζί της, όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι ήταν αρκετά επικοδομητική, τουλάχιστον για τη δική μου ομάδα, τους σοσιαλιστές. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να καταλήξουμε σε κάτι χρήσιμο. Το το χρήσιμο αυτό πρέπει να είναι επωφελές βέβαια και για τους καταναλωτές. η εισαγωγή της τεχνολογίας, της και, της, ε, τεχνολογίας και, της, ε, και των επικοινωνιών, ε, η κινητή τηλεφωνία είναι κάτι το οποίο έζησε η δική μας γενεά και θα σημαδέψει ακόμα περισσότερο τις επόμενες γενναίες. Υπάρχουν βέβαια διαφορές ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ε, ε, έχουν αρχίσει να μειώνονται όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες. Παρόλα αυτά, αυτός ο νέος τομέας που είναι πολύ συναρπαστικός για τους καταναλωτές είναι δύσκολος ε, για τους ε, ε, παρόχους γιατί η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει 120 με 130 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι πιο σημαντικό το, είναι πιο σημαντική απόδοση της κινητής τηλεφωνίας από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιο είδους ρύθμιση, γιατί είναι απαραίτητο μάλιστα, γιατί διαπιστώσαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Μάλιστα, όταν οι, οι καταναλωτές μας έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ε, ε, φοβερή ε, νέα τιμολόγηση, την πολύ δαπανηρή, όταν πρέπει ας πούμε να τηλεφωνήσει ή και να του τηλεφωνήσουν και ούτως ή άλλως να πληρώνει. Είτε του τηλεφωνούν είτε τηλεφωνεί. Ή όταν και αυτός που τηλεφωνεί και αυτός τον οποίο τηλεφωνούν πρέπει και οι δύο να πληρώσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές ε, πολύ υψηλούς λογαριασμούς, διωγγωμένους, ειδικότερα για τους ε, ε, καταναλωτές που ταξιδεύουν πολύ, που μετακινούνται πολύ και καταλήγουμε σε γελίες καταστάσεις, Δηλαδή πολλές φορές οι τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές ε, από το Αμβούργο στο Μόναχο ή από το Μόναχο ε, στη Βαβαρία. Όλες παρόλες τις προσπάθειες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθεί η υπερβολική αυτή τιμολόγηση, τα πράγματα παραμένουν ακόμη πολύ δύσκολα. Λιγότερο από 4% των ε, κλίσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησαν σε τζίρο 5 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ για τους παρόχους και μιλάω για τους τελευταίους αριθμούς που έχω υπόψη μου. 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για να μπορέσουμε να ε, παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες ε, στους καταναλωτές και καταλήγουμε σε τεράστια ποσά για μια υπηρεσία η οποία είναι μια πολύ μικρή περιορισμένη υπηρεσία που, που προσφέρουν ουσιαστικά οι πάροχοι. 80% της ε, αγοράς ε, ανήκει σε τέσσερις μεγάλους ε, παρόχους. Είμαστε λοιπόν περίπου σε κατάσταση καρτέλ, όπως το είχε πει και ο συνάδελφος Charles Chichester και τον παραθέτω εδώ οι οποίοι αντιστέκονται ε, στα διαρθρωτικά μέτρα και τα, ε, τις τιμολογήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς θα χρειαστεί επομένως ε, σε, στο προβλέψιμο μέλλον να ρυθμίσουμε με κάποιο τρόπο αυτό το, την αγορά της περιαγωγής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα λοιπόν ότι τέσσερις ε, μεγάλες εταιρείες μοιράζονται το 80% της αγοράς. Μιλάμε δηλαδή για εταιρείες ε, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται λοιπόν, είναι παρούσες σε όλες τις χώρες, είτε οι ίδιοι είτε σε συνεργασίες με τους, με, με τους εθνικούς παρόχους. Οι τέσσερις αυτοί ε, πάροχοι ε, θεωρητικά διατηρούν τα εθνικά ε, σύνορα μόνο για λόγους τιμολόγησης, για να μπορούν δηλαδή να χρεώνουν παραπάνω. Ενώ εκείνοι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά διαχειρίζονται ολόκληρο το σύστημα. Ή αν έχουν πραγματικά αν έχουμε πραγματικά μία ενιαία αγορά και στοχεύσουμε σε μία ευρωπαϊκή αγορά ε, της τηλεφωνίας, θα μπορέσουμε να υπερβούμε αυτό το πρόβλημα της ε, της περιαγωγής, ελπίζω μέχρι το 2015. Εγώ, έτσι λέω εγώ, αλλά αν μπορέσουμε και νωρίτερα, ακόμη καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα που θέτει η Αγγέλικα Νίβλερ, εμείς είμαστε υπέρ των διαρθωτικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως μόνο προσωρινά. Γιατί ο τελικός μας στόχο πρέπει να είναι μία ε, ενιαία τιμολόγηση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε με το local breakout όπως ε, αναφέρεται στη συμβιβαστική τροπολογία της ε, Δεν μας ε, ικανοποιεί πάρα πολύ αυτή η ρήτρα μη συμμετοχη opt ε, opt-out για κάποιους ε, φορείς που στόχο έχει να εχμαλωτίζει τον πελάτη. σε μία φυλακή τον καθυλώνει και δεν του επιτρέπει να κάνει και καμία επιλογή. Ούτε του επιτρέπει να υποφελείται από χαμηλότερες τιμές. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ της ε, ενιαίας ευρωπαϊκής ε, τιμολόγησης. Κάτι τέτοιο όμως ε, λέγεται ότι δεν θα επιτρέπει τον ανταγωνισμό των φορέων. Όταν βλέπω την έλλειψη ανταγωνισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εγώ θα προτιμούσα να αναλάβω αυτό το, το ρίσκο, αρκεί να καταφέρουμε να υπερβούμε το πρόβλημα της περιαγωγής και να ε, έχουμε κάποιες λογικές τιμές, εν πάση περιπτώσει, σε όλες τις 28, 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκέμπελς. Η κυρία Βαλεάν από τους Φιλελευθέρους, σας παρακαλώ πέντε λεπτά αν μπορείτε να μιλήσετε. Αρκούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς κυρία Νίμπλερ σας ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο των συμβιβαστικών τροπάσεων που προτείνατε και το γεγονός ότι ήσασταν διατεθειμένοι να συμπεριλάβετε τις διάφορες συναλλακτικές λύσεις που σας προτείναμε. Εχθέ είχαμε αυτή τη συνεδρίαση μαζί σα και με τους κοιόδης συζητητέ. παρά το γεγονός ότι για μένα ήταν πολύ επικοδομητική. Μέχρι το τέλος τη συνεδρίασης εξακολουθούσα να πιστεύω ότι δεν έχουμε μία απόλυτα ορθή λύση για το θέμα της περιαγωγή, Διότι τώρα εξετάζουμε μία διαρθρωτική λύση και αυτό για ποιο λόγο, γιατί θέλουμε να υποχρεώσουμε τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή έχουμε ανταγωνισμό στις ε, διεθνείς αγορές ε, και η περιαγωγή ξεκίνησε σαν ε, μια υπηρεσία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Με στόχο όμως αυτό, το να υποβοηθήσουμε τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Νομίζω ότι τελικώς δεν διασφαλίζουμε ότι υπάρχει σαφές όριο μεταξύ τιμών, ε, ανώτατων τιμών χονδρικής και λιανικής ε, και έτσι δημιουργούμε πρόβλημα στην αγορά. Και παρά το γεγονός ότι δεν ήμουν διατεθειμένη να ε, αγγίξω τις τιμές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ξεκινάει η συζήτηση για τις τιμές ε, θα προκύψουν πάρα πολλές ιδέες και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ομάδα μου θα ήθελε μια συμβιβαστική πρόταση για τις τιμές υπό τον όρο να μπορέσουμε από κοινού να βρούμε κάποια κριτήρια για να καθορίσουμε τα ανώτατα όρια τιμών. Παραδείγματο χάρη, θεωρώ ότι το περιθώριο για τις νέες εισόδους θα πρέπει να είναι αυτό που προτείνεται από τον κύριο Μπέρεκ ε, με την μέθοδο υπολογισμού που υπολογίζει στα 2 τρίτα ε, και χωρίζει σε 3 τρίτα τα εισόλες ανώτατες τιμές και θα ήθελα να υπολογιστούν οι τιμές με αυτόν τον τύπο. Δεύτερον, πρότεινα επίσης να επεκταθεί το ανώτατο όριο μέχρι το 2015 ώστε σε κάποιες περιπτώσεις να μπορούμε να έχουμε και τα ανώτατα όρια που προτείνονται από την κυρία Νίμπλερ, αλλά και να μπορέσουμε να αναβάλουμε την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2016, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά και ε, ίσως να αποφασίσουμε να επεκτείνουμε τον κανονισμό για να υποβοηθήσουμε τον ανταγωνισμό. Με χαρά βέβαια διαπιστώνω ότι και η συγγήτρια είναι προς την ίδια άγουσα ε, ως προς την ε, συμβιβαστική τροπολογία για τα ανώτατα όρια. Θα ήθελα επίσης ε, να χαιρετήσω την εισαγωγή αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης δύο χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του κανονισμού. Όσον αφορά τώρα το local breakout, σας είμαι ευγνώμων διότι το είχα προτείνει εγώ και βλέπω ότι το δέχεται η συγγήτρια στη συμβαστική της τροπολογία και από ό,τι φαίνεται το υποστηρίζουν ευρύτατα ε, ε, τα μέλη της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι το local breakout συμπληρώνει τα διαρθρωτικά μέτρα και κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό ε, να μειώσουμε τις τιμές μεταφοράς δεδομένων, ε, διότι γίνεται μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Παρά το γεγονό ότι δεν είναι περιαγωγή αυτή καθε αυτή, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά στον κανονισμό κατά με. Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 4α υπάρχει μία διάταξη που ε, δεν επιτρέπει στους πελέτες να έχουν εναλλακτικό συμβόλαιο σε αυτή την περίπτωση και αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα του opt-out θα πρέπει οι πελάτες που έχουν εναλλακτικό συμβόλαιο να μπορούν να υποφαληθούν από την συμπληρωματική λύση του local breakout. Όσον αφορά τώρα τη ρήτρα τη συμπληρωματική που έχουμε στο άρθρο 4, παράγραφος 8 νέα στη συμβιβαστική πρόταση, θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για την εφαρμογή της, αυτό το σύστημα της καταποκοπήν ε, χρέωσης είναι πολύ πιο φιλικό προς το χρήση και πολύ πιο απλό. Και επίσης ε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να απαντήσει και στο στόχο μας, δηλαδή να μειώσουμε τις τιμές της περιαγωγής και να φτάσουν στις τιμές ε, της εγχώριας τιμολόγησης ανάλογα με την κάθε χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει αυτή η ρήτρα opt-out παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αποφασιστούν για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Επί έστω ότι έχουμε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ας πούμε από τη Ρουμανία, που να μπορεί να προσφέρει φθηνότερες ε, συμφωνίες περιαγωγής από έναν ε, Βέλγο, μια βέλγικη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να ενταχθεί στην ε, βελγική αγορά, ακόμα και αν προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία, αλλά κατ' εμέ θα ήταν μια καλή λύση. Όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι ε, η Μπέρεκ θα πρέπει να αποφασίσει ποιος είναι ο ορισμός των τιμών περιαγωγής ε, και να είναι σχεδόν ισότιμες με τις εγχώριες τιμές, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο επί του ζητήματος, διότι πρόκειται για μια πρόταση η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι παρέμβαση και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε με ένα διαρθρωτικό μέτρο. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτ. Ε, ε, για να εξοικονομήσω χρόνο δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκέμπελτ γιατί για μια φορά συμφωνώ 100% με ό,τι είπε όσον αφορά τη χρυσομένη φυλακή είναι μάλλον για τον πάροχο και όχι τόσο για τον πελάτη όσον αφορά την ε, μεταφορά δεδομένων και την τιμολόγησή τους νομίζω ότι είναι 500 ευρώ ανά γιγαμπάιτ δηλαδή σε αυτή την επιτροπή πολύ συχνά ακούω ότι θέλουμε να αναπτύξουμε την διακίνηση του ίντερνετ ε, αλλά με αυτές τις τιμές δεν θα το επιτύχουμε οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν σχετικά με την διακίνηση των δεδομένων ε, και ξέρω ότι πολλοί σκιώδεις εισηγητές έχουν κάνει μια πανεφερή πρόταση και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο διότι από την ε, οπτική γωνία του ε, καταναλωτή θα μας κοροϊδέψουν διότι θα, ή θα θεωρήσουν ότι τους κοροϊδεύουμε εμείς. Επίσης, ε, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο στόχος μας, ε, διότι αν ε, κάποιος δίνει τιμές περιαγωγής ε, ε, ίδιες ε, με το εσωτερικό της χώρας γιατί θα προσπαθήσει να βρει ο πελάτης κάποιον καλύτερο. Εάν λοιπόν ζητήσουμε να υπάρχει πλήρης ελευθερία για τους καταναλωτές οι δυνάμεις αγοράς θα υποχρεώσουν τους παρόχους να ευθυγραμμίσουν τις τιμές περιαγωγής με τις τιμές στο εξωτερικό στο εσωτερικό. Ε, πιστεύω ότι το βασικό είναι να υπάρχει ένα πλαφόν στις τιμές. Ξέρω ότι δεν είναι τέλεια η λύση μας, αλλά κανείς δεν έχει βρει την ε, τέλεια λύση και γι' αυτό συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε λήψη μιας καλύτερης λύσης. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Όχι, δεν θα παρέμβει, άρα τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις. Η κυρία Δελκαστήγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ τη συνάδελφο Νίμπλερ, διότι διαχειρίζεται και καθοδηγεί το θέμα αυτό με εξαιρετικό τρόπο ε, έχει λάβει τη σωστή άγουσα και κατ' εμέ έχει και μία στάση που θέλει να συμπεριλάβει τα πάντα, βέβαια πάντα με ε, γνώμονα τι είναι αποτελεσματικό, διότι αν είναι κάτι μη αποτελεσματικό δεν αξίζει. Θα σταθώ στο ανώτατο όριο, εκεί τελείωσε ο συνάδελφος Φίλιπ Λάμπερτ και νομίζω ότι είμαι βέβαιη ότι θα ακουστεί και κάποιο άλλος προ την ίδια κατεύθυνση, ότι δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η ρήτρα opt-out, διότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις ε, προηγούμενες ε, διατάξεις για την περιαγωγή γίνεται για να γίνει παρέμβαση ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της αγοράς περιαγωγής, διότι στην πραγματικότητα η δράση μας ε, καθορίζει τις δυνατότητες επιλογής των χρηστών μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα βήμα παραπάνω και θέλει να ανοίξει την αγορά δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν περισσότεροι ανταγωνιστές αλλά και ο τελικός στόχος είναι να υπάρχουν καλύτερες επιλογές και καλύτερες τιμές για τους χρήστες. Υπάρχουν όμως πιο άμεση και πιο έμεση τρόποι και πιο ευέλικτοι τρόποι για να επιτύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ αυτής της ε, ελεύθερης επιλογής των καταναλωτών, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα στην κατάσταση την οποία ε, ζούμε βάσει αυτής της νέας νομοθεσίας, στην οποία θέτουμε ε, όρους για την ε, χρήση αυτής της αγοράς και τελικώς για τους τελικούς χρήστες αυτής της αγοράς, ε, δεν ε, δίνουμε τη σωστή κατεύθυνση και κατ' εμέ νομίζω ότι δεν είναι ενδιαφέρον να υπάρχει το opting out, διότι το opting out σημαίνει ότι τελικά πιέζουμε κάποιον να κάνει καλύτερες τιμές, όπως είχαμε προβλέψει με τα ανώτατα όρια. Πιέζουμε λοιπόν να υπάρχουν καλύτερες τιμές, διότι δίνονται κίνητρα στους ε, εγχώριους παρόχους να δίνουν καλύτερες τιμές ε, στους πελάτες τους για τις ε, τιμές περιαγωγής. Εάν λοιπόν ένας καταναλωτής ε, κάνει μια συμφωνία με την εταιρεία κινητής του τηλεφωνία για να έχει κάποιες τιμολογήσεις οι οποίες ουσιαστικά θα είναι ισοδύναμες με τις εγχώριες τιμές, ίσως είναι λογικό να μην εφαρμόζεται η ρήτρα η οποία θα υποχρεώνει να έχει κάποιος ε, μία, ένα πάροχο μόνο για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Τώρα, θα πρέπει βέβαια να δούμε τι σημαίνει αυτό το ισοδύναμο, διότι το ισοδύναμο μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος με διαφορετικό τρόπο. Και εγώ στην τροπολογία μου ε, το πρότεινα κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να επισέλθει η Μπέρεκ, ο φορέας των ρυθμιστών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος θα δώσει το ε, τη γνωμοδότησή του και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη γνωμοδότηση της Μπέρεκ θα πρέπει να αποφασίσει αν η τιμή που προσφέρει ε, ο εγχώριος πάραχος και δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και τι γίνεται με αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ισοδύναμη ή όχι, αν είναι δηλαδή πρακτικά ισοδύναμη ή όχι και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογή από πλευράς Μπέρεκ. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να έχουμε τη ρήτρα του opting out με τις απαιτήσει που έχω θέσει όμως. Ευχαριστώ κύριο Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκλογή σας και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι ξαναβρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή στην οποία ήμουν και στην προηγούμενη θητεία και ελπίζω να μπορέσω να συνεισφέρω και να έχουμε και μεγάλη συνέργεια με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ιδίως για τα θέματα ενέργειας. Questo αυτό ε, σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να συνεισφέρω πολύ θετικά στο θέμα αυτό. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ όμως την κυρία Νίμπλερ για την παρουσίαση που μας έκανε και θα ήθελα να συνεχίσω από την παρέμβαση που είχα κάνει στην προηγούμενη επιτροπή Θεωρώ ότι η συμφωνία με τον... Ε, εδώ συμφωνώ με τον κύριο Γκέμπελς ότι το roaming είναι μια παράλογη λύση. Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας μπορούν αυτή τη στιγμή να παρουσιαστούν στον ε, καταναλωτή ως ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις με συνεργασία μεταξύ τους και με τη δυνατότητα να θεωρούν την Ευρώπη ως νέα αγορά. προσεγγίζουμε μεν το στόχο, αλλά πόρο απέχουμε και ταυτόχρονα. Ίσως την επόμενη φορά που θα το συζητήσουμε, να μπορέσουμε στην πράξη να πείσουμε τις επιχειρήσεις να παρουσιάζονται στο χρήστη ως μία μοναδική μεγάλη υπηρεσία ε, για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόντι, Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για τον ορισμό σας. Έκανα εντατικά Ιταλικών, ελπίζω ε, στο μέλλον να είστε ε, μαζί μου. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Νίμπλερ για την έκθεσή της, ε, γιατί παίρνει, κάνει ένα βήμα μπροστά και βλέπει περισσότερο προς το μέλλον, όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για τους διάφορους, ε, διάφορους συμβιβαστικά κείμενα. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, τι θα πει η περιαγωγή, είναι κάτι το παροχημένο. Πολύ παροχημένο, μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο 2012 είναι ο πιο ε, γρήγορα μεταβαλλόμενος τομέας της ε, τεχνολογίας. Ε, δεν είναι επαρκή αυτά που κάνουμε μακροπρόθεσμα. Έχουμε μία νέα πολιτική φάσματο, θα επανέλθουμε και στο μέλλον και μακροπρόθεσμα θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόκληση για τους παρόχους ήδη σήμερα. Όμως... Θα ήθελα κάτι ακόμη να επισημάνω. Και αυτό είναι ότι ο όγκος ε, της ε, κυκλοφορίας ε, δεδομένων αυτό είναι το βασικότερο, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ε, τα δεδομένα ε, μετακινούνται με όγκους όλο ένα και αυξανόμενους, ε, διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ο όγκος τους ε, ε, κάθε χρόνο και αν δούμε τους τελευταί, τα τελευταία πέντε χρόνια νομίζω ότι έχει δεκαπλασιαστεί μάλιστα. Και αυτή τη χρονιά πάλι θα διπλασιαστεί και κάθε νέα γενεά ε, έξυπνου κινητού ε, ή ηλεκτρονικού υπολογιστή συμπεριλαμβάνει νέες υπηρεσίες. Πριν από δύο χρόνια ο, η λέξη app, εφαρμογή, ε, δεν ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Σήμερα όμως η λέξη αυτή ουσιαστικά, ουσιαστικά συμβολίζει τον αριθμό των νέων υπηρεσιών. Όλο και περισσότερες ε, εφαρμογές υπάρχουν, ε, όλο και πιο χρήσιμες είναι και κάθε γενεά iPhone σημαίνει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. Μπορεί βεβαίως να πούμε ότι θα μειώσουμε τα ανώτατα όρια των τιμών αυτό δεν αρκεί όμως. Ε, αν ο όγκος των δεδομένων τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, τότε το το 2014 είναι πολύ μακριά αν έχουμε πολλαπλασιασμό κάθε χρόνο. Επομένως πρέπει να ε, αλλάξουμε τις παλιές μας ε, στρατηγικές και συμφωνώ με την κυρία Νίμπλερ ως προς αυτό. Και αυτό μας θα πρέπει να είναι και το πρώτο μας βήμα. Δεν βλέπω κανένα επιχείρημα. Έχω ακούσει παρόχους ε, να λένε ότι δεν ε, ε, τους αρέσει το σύστημα που προτείνεται γιατί θεωρούν ότι οι υπόλοιποι πάροχοι θα υποφεληθούν και όχι οι ίδιοι. Όμως αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα κατά, είναι ένα επιχείρημα υπέρ του συστήματος, γιατί έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Και από τεχνικής απόψεως αυτό που θα σημαίνει είναι ότι θα καταφέρουμε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το τοπικό δίκτυο με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Wi-Fi, το ασύρματο ε, ε, δίκτυο, ε, εδώ μέσα ή στο ξενοδοχείο μας για παράδειγμα. Θα λύσουμε και το πρόβλημα με τα γραπτά μηνύματα, τα SMS και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ως γνώμονα για την νομοθεσία γιατί όλα τα υπόλοιπα μετά θα ακολουθήσουν να λύσουμε αυτό το βασικό πρόβλημα. Αν ο κύριος Λάμπερτ μπορεί να συμφωνήσει 100% με τον κύριο Κέμπελς, εγώ μπορώ ε, κατά 10% τουλάχιστον να συμφωνήσω μαζί του είναι γεγονός ότι οι τοπικοί ε, παροχοί θα έχουν πάντοτε τους υψηλό, τις υψηλότερες τιμές. Και αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε αυτό το breakout. Γιατί τότε ένα από τα, προβλήματα, ε, τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε θα ε, επιληθούν και θα είναι πιο δυναμικό το σύστημα. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ την κυρία Νίμπλερ για την έκθεσή της. Grazie, la parola al collega ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο τώρα. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Αγγέλικα για την ε, ε, προεργασία και πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε ότι η κινητή τηλεφωνία έχει όλο και μεγαλύτερο ο κύκλο εργασιών και κέρδη αλλά και δημιουργεί και περισσότερες θέσεις εργασίας. Πάντοτε λοιπόν έχουμε τονίσει ότι οι τηλεπικοινωνίες πρέπει να επενδύουν για να έχουμε νέα δίκτυα και νέες τεχνολογίες. Τρίτη παρατήρηση. Στις εθνικές αγορές έχει εξελιχθεί μια εξαιρετη... ένας εξαιρετικός εσωτερικός ανταγωνισμός. Είναι εξαιρετική εξέλιξη και έχουμε μόνο ένα πρόβλημα στο roaming στην περιαγωγή και προσπαθήσαμε να το λύσουμε με μία από μονοκονδυλιά. Βέβαια μειωθήκαν οι τιμές αλλά δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός και άρα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη σωστή λύση για τον ανταγωνισμό και πρέπει τώρα η κατάσταση να χαλαρώσει για να μπορούμε να επιτύχουμε στην το ίδιο το οποίο έχουμε και σε εθνικές αγορές. Πιο έντονος ανταγωνισμός. Ο καθένας να μπορεί να επιλέγει μέσω ποιου θα επικοινωνεί και θα τηλεφωνάει. Γι' αυτό και θα έπρεπε να στηρίξουμε την Αγγέλικα να ε, προχωρήσουμε γρήγορα σε διαρθρωτικές αλλαγές και δεύτερο να μην καθορίσουμε τις τιμές γιατί ε, ε, πάμε αντίθετα στην εξέλιξη που επιζητούμε. Δεν πρέπει λοιπόν να απελευθερώνουμε από τη μία μεριά και να περιορίζουμε από την άλλη. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν την ε, ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ας μην επικεντρωθούμε τόσο πολύ στον καθορισμό τιμών. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ μπορώ να, σας, να συμφωνήσω και να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό με μέτρα και πώς θα πιέσουμε την αγορά. Διότι παραδείγματο χάρη υπάρχει η ιδέα opt-out, η ρήτρα αυτή που είναι μια καλή ιδέα ε, γιατί τότε ο πάροχος θα ε, ε, επενδύσει σε περισσότερη τεχνική διότι διαφορετικά δεν θα έχουμε τα σωστά μέτρα. Το local breakout είναι και αυτό μία δυνατότητα για να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άκουσα και μία ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία μπορεί να προωθηθεί μέσω ενός αριθμού ε, πανευρωπαϊκού που θα προεπιλόγουμε αλλά δεν θα ήταν ευλακώδες να πούμε ότι η Ευρώπη θα έχει έναν ενιαίο αριθμό προεπιλογής για να λύσουμε το πρόβλημα αλλά κύριε Ρόιλ έχετε δίκιο αυτό πρέπει να σκεφτούμε εδώ είναι ότι αν ρίξουμε πολλές τις τιμές δεν θα έχουμε νέους παρόχους στην αγορά και το πρόβλημα αυτό θα υπάρχει και το πρόβλημα της αγοράς είναι το πρόβλημα των μεγάλων που έχουν τα δίκτυα, που έχουν τις γραμμές και αυτοί μπορούν να κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις και οι μικροί δεν μπορούν να κάνουν τόσες προσφορές Θέλουμε λοιπόν ε, να βρούμε ε, λύσεις ε, μέσω της οικονομίας της αγοράς για να μπορέσουμε να εντείνουμε τον ανταγωνισμό και γι' αυτό κυρία Νίτλερ όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι είμαστε υπέρ του opt-out και του local breakout και ε, τώρα αρχίζει το παζάρι, θα υπάρξει και μία σκιώδης έκθεση, αύριο θα υπάρχουν συνεδριάσεις των σκιωδών ε, εισηγητών και θα παρακολουθήσω το θέμα αυτό μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ρούμπικ, ε, θα ήθελα να ρωτήσω και αν έχετε και τις κάρτες ε, για να ψηφίσουμε στη συνέχεια. Κύριε Ρούμπικ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βεβαίως και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν πρέπει να καθορίσει τιμές. Αυτές πρέπει να διαμορφώνονται μέσω του ανταγωνισμού. Αλλά αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε είναι να καθορίσουμε που υπάρχει παραβίαση και ξεκινά και είναι το σημείο που ξεκινά η παραβίαση διότι παραδείγματο χάρη στη χώρα μου υπάρχει ένα πακέτο ο, χίλια λεπτά, χίλια SMS, ένα ε, gigabyte και κοστίζει 8,8 ευρώ. Εάν όμως έρθω στο Βέλγιο ενδέχεται το ένα ε, gigabyte να μου κοστίσει 13.000 ευρώ και εμεί θέλουμε να καθορίσουμε τα 500 ευρώ σαν όριο. Οπότε ε, θέλουμε να υπάρχει ένα όριο να μην ξεπερνάει κανείς και να μην παραβαίνει τα 500 ε, ευρώ ενώ στη Γερμανία είμαστε στο 8,80 ευρώ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν τεχνικές διορθώσεις για να υπάρξει αληθινός ανταγωνισμός γιατί βλέπουμε ότι σε, νέ, ε, σε πολλές νέες τεχνολογίες ε, ε, όπου έχουμε όλους τους Ευρωπαίους που διακινούνται ΙΟΣ θα πρέπει πάνω από 90 εκατομμύρια θα πρέπει ε, να υπάρξει ένας καθορισμός τιμών ο οποίος να είναι εφικτός και ρεαλιστικός. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από εμάς για την ανάληψη της Προεδρίας ε, της Επιτροπής Ήτρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και τη σημερινή συζήτηση και από ό,τι φαίνεται είναι δεσμευμένοι όλοι ενδιαφερόμενοι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για να υπάρξει συμφωνία για την περιαγωγή πριν εκπνεύσει η παρούσα συμφωνία τον Ιούνιο. Ε, μας ενθαρρύνει η προσέγγισή σας για τις συμβιβαστικέ προτάσεις και θα θέλαμε να συγχαρούμε το Κοινοβούλιο για την επικοδομητική του προσέγγιση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και από πλευρά μας για να επιτύχουμε αυτό τον κοινό στόχο. Ε, γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα και θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε για να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Ε, με χαρά πρέπει να σας πω ότι προχωρούν και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο με επικοδομητικό τρόπο και ακούσαμε και τις συζητήσεις σας εδώ σήμερα στην Επιτροπή Ήτρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσας, ε, πολύ σημαντική συζήτηση για μας και αποδεικνύει ότι οι ανησυχίες και οι προκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανάλογες με αυτές του Συμβουλίου και προσβλέπουμε ε, στην ανάλυση των συμβιβαστικών προτάσεων όταν θα τις λάβουμε για να προετοιμάσουμε και τον διάλογό μας. Σας ευχαριστώ προς το παρόν και προσβλέπουμε στην ε, καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εάν συμφωνούν και οι συνάδελφοι, θα διακόψουμε τώρα για την ψηφοφορία και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά την ε, ψηφοφορία. Ο κύριος Γκέμπελς. Euh, Μία μικρή παρατηρήση, κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Ρούμπικ είπε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να ε, μπει στη διαδικασία του ορισμού των ε, τιμών. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, χωρίς τον κανονισμό περιεγωγή 1 και περιεγωγή 2, στον οποίο Ακριβώς το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο παρενέβησαν, δεν θα είχαμε φτάσει πουθενά, γιατί ο ανταγωνισμός δεν θα είχε οδηγήσει σε στη μείωση τιμών που ήθελε το Κοινοβούλιο. Ναι συνάδελφοι, θα ήθελα όμως να τονίσω ότι και εγώ είμαι υπέρ των περιορισμών, δηλαδή να μην μπορεί κανείς να κάνει καταχρήσεις, αλλά δεν θέλουμε το Κοινοβούλιο να καθορίσει μία ενιαία τιμή και να πούμε ένα gigabyte, ένα ευρώ και αυτό να είναι το μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των φθηνότερων και των πιο ποιοτικών και ε, θα μειώσουμε όμως κατά το ίμιση της τιμή ε, τότε δεν ξέρουμε ε, πώς θα γυρίσει κανείς προς τα πίσω αν χρειαστεί. Εδώ κάνουμε μία εξαίρεση για τις τηλεπικοινωνίες διότι υπήρχαν πάρα πολύ ψηλές τιμές αλλά επειδή ήμουν ο διαπραγματευτής για το roaming 1 και 2 για το ΕΛΚ ξέρω ακριβώς ε, πώς τα καταφέραμε. Ωραία, ευχαριστώ. Διακόπτε τη συζήτηση. Θα συνεχιστεί αμέσω μετά την ψηφοφορία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Λίμπλερ για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Ε, λογικά θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Ξεκινούμε με την έκθεση της ε, συναδέλφου Χοκμάρκ. Ε, μία ψήφο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρασης ψηφοφορίας. Έχουμε δύο μέλη από το ΕΛΚ επιπλέον. Δύο αναπληρωτές σας παρακαλώ να βγάλετε το καρτιλάκι σας. Η κυρία Χολ. Νομίζω ότι δεν δουλεύει το μηχάνημά μου, λέει η κυρία Χολ. Μπορεί κάποιος να δει τι γίνεται με τη συσκευή της κυρίας Χολ που δεν δουλεύει ή αλλάξτε θέση ένα λεπτό να ψηφίσουμε. Ωραία. Άρχεται και πάλι ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, ξέχασα την κάρτα μου στο Στρασβούργο. Δύο συνάδελφοι λοιπόν ψηφίζουν χωρίς κάρτα και υπερψηφίζουν. Δύο συνάδελφοι λοιπόν ψηφίζουν υπέρ. Υπάρχει ακόμα ένα μέλος από το ΕΛΚ επιπλέον. Ωραία. πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 52 ψήφους υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Απόλυτη ομοφωνία. Να περάσουμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία. Έκθεση Γιώχανσον Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1α σημείο 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την ε, τροπολογία 6 της παραγράφου 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας, 29 ψήφοι υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1α, τροπολογία 7 της κυρίας Τσικάου, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1, 8. Τσικάου, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Η τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 33, μπουτικόφερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 παράγραφος 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Της κυρίας Τσικάου κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38, παράγραφος 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία για την τροπολογία 41 του κυρίου Μπουτικόφερ. Συμφωνούν όλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 τσουκαλάς υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4, 45, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Παράγραφος 4, 46, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, 48, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Α, με συγχωρείτε. Ξέχασα την τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, όχι, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 55. Τρία μέλη του ΕΛΚ επιπλέον. Δύο επιπλέον. Ένας επιπλέον. Ένας φιλελεύθερος επιπλέον. Ωραία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πενήντα επτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πενήντα οκτώ Κάριν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 Φράνκο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 59. Check sul 59. Και πάλι ένα επιπλέον από το ΕΛΚ. Ένα επιπλέον από το ΕΛΚ. Sorry. Maybe I created them. Ε, συγγνώμη, μάλλον δημιουργήσα κάποια παρανόηση. Νομίζω ότι το δεύτερο τμήμα της 58 δεν εγκρίθηκε και θα ήθελα να αμφισβητήσω το αποτέλεσμα αυτό. Και είχατε δίκιο εσείς, ναι. Λοιπόν, εγκρίναμε. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Εγώ φταίω. Δεν έθεσα προς ψήφιση το δεύτερο τμήμα της 58. Επομένως, την 59 την εγκρίνουμε. Μπορούμε να ε, ψηφίσουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της 58. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Ο κύριος Φράνκο, παρακαλώ. Προτείνω το Ask for Financial Instrument να το διαγράψουμε για να είναι πιο συνεκτικό το κείμενο. Διακόπτη, Πρόεδρος. Συγγνώμη, συζητάμε την 60. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 58. Κύριε Δελκαστήγιο. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Δελκαστήγιο. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Για να ακολουθήσουμε τον κατάλογο του ΕΛΚ για το πρώτο τμήμα υπάρχει ένα συν, αλλά για το δεύτερο τμήμα για την τροπολογία του αγαπητού συναδέλφου υπάρχει ένα πλήν που πρότεινε ο σκιώδης συζητητής. Έχουμε πλήν για την ψηφοφορία του ΕΛΚ βάσει του καταλόγου ψηφοφορίας για το δεύτερο τμήμα της 58. Ωραία, ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ψηφίζουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 58, παράγραφος 5, υπέρ. Κατά. Κατά την άποψή μου απορρίπτεται. Αν θέλετε μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Βότο απέρτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 20 ψήφοι υπέρ, 31 κατά. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 60 και να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Φρανκ προτείνω να διαγράψουμε το Ask for Financial Instruments για να είναι πιο συνενετική η πρόταση και ε, επιτρέπει για μεγαλύτερη ευελιξία. Δέχεστε την πρόταση του κύριου Φράγκο. Καλώς. Ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 60 ως τροποποιήθηκε από τον συνάδελφο Φράνκο με τη διαγραφή ε, της φράσης υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 τσικάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 βαμπρέμπ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 665 του συνάδελφου Ρόιλ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 βαμπρέντ, υπέρ. ξεχνώ συνέχεια το δεύτερο τμήμα. Πρέπει να το μάθω. Ζητώ συγγνώμη. Θα μάθω, θα μάθω. Δεύτερο τμήμα λοιπόν του 65. Όχι. Όχι, συγγνώμη. Ο κατάλογος που έχω εγώ εδώ Συγγνώμη, ο κατάλογος μου λέει ότι το πρώτο τμήμα καταπίπτει αν ε, εγκριθεί η συμβαστική τροπολογία 8, η οποία και εγκρίθηκε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν καταπίπτει. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Ναι, βεβαίως. Εγώ είχα μόνο ένα τμήμα το οποίο έπρεπε να υποβάλω σε ψήφιση που ήταν το δεύτερο τμήμα. Επομένως, ε, ξέχασα να σας πω ότι ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Το πρώτο είχε ήδη διαγραφεί από τον κατάλογό μου και επομένως Ξαναψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 65 ε, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 μπουτικόφερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 μπουτικόφερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική κλίση το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας επιπλέον από το ΕΛΚ. Εξαιρετικά. Έχουμε και δύο επιπλέον ψήφους υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν με 51 ψήφους συν 2, 53 ψήφους υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά, συγχαρητήρια. Ζητώ συγγνώμη για τα μικρά μου λαθάκια, σας υπόσχομαι ότι θα μάθω. Και να επανέλθουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Να περιμένουμε να αποχωρήσουν αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Ε,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 Παρακαλώ, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ε, σα συγχαρώ καταρχά ε, εσάς ε, για το νέο σας ρόλο ω, πρόεδρο της Επιτροπής και να συγχαρώ και την κυρία Νίμπλερ για την εξαιρετική τη εργασία για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, φιλοδοξία της ε, Επιτροπής σας για την περιαγωγή, ώστε να ληφθεί σύντομα μία απόφαση για να μην υπάρχει κενό μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης συμφωνίας. Η κυρία Νίμπλερ έθεσε μερικά ζητήματα στην αρχή, δεν αποτελεί έκπληξη. Το είχα θέσει και εγώ το ζήτημα αυτό πολλές φορές ε, στην Επιτροπή σας. Ε, ε, όταν εξετάζουμε την πρόταση και τις διαφορές των τιμών, δεν θα πρέπει να τα δούμε απομονωμένα από την υπόλοιπη πρόταση και ειδικότερα από τα διαρθρωτικά μέτρα. Πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό που είπε ο κύριος Κρόιτσμαν και η κυρία Βαλεάν, ότι πρέπει να αφήσουμε επαρκές περιθώριο μεταξύ των τιμών χονδρικής και λιανικής, ώστε να υπάρχει και κίνητρο αλλά και περιθώριο για τους ε, ε, νέους ε, παίκτες της αγοράς και βέβαια να υπάρχει όφελος και για τους πελάτες της περιαγωγής. Όταν συζητούμε λοιπόν τις διαφορές των τιμών Ενδεχομένω να υπάρχει περιθώριο να επανεξετάσουμε ποιο είναι το ε, σωστό ανώτατο όριο χονδρικών τιμών, αλλά πρέπει να επιτρέψουμε και ένα ασφαλές περιθώριο μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής. Όσον αφορά τώρα ε, τις τιμές ε, περιαγωγής δεδομένων ε, που εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλές, ειδικότερα για κάποιον που χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα, ακόμη και με, τα, με τις τιμές που, προτείνονται, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την λύση για το local breakout, ε, οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο των ε, ε, ανώτατων ορίων για τα δεδομένα, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της περιαγωγής δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε νέες καινοτόμε λύσεις και είναι γεγονός ότι το local breakout θεωρείται μια πάρα πολύ καλή λύση. Εμείς θα το εξετάσουμε και ελπίζουμε να ενισχυθεί και ο ανταγωνισμός, ειδικότερα όσον αφορά τα ε, δεδομένα. Τώρα όσον αφορά την ρήτρα opt-out. Ε, είναι πράγματι πολύ ελκυστική η πρόταση και είναι σαν να μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα με μια μαγική ρήτρα που θα τη συμπεριλάβουμε ε, στην πρόταση, αλλά πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι υπάρχουν ενδεχομένως και αρνητικές συνέπειες της πρότασης αυτής. Δηλαδή, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μια τέτοια ρήτρα υπόκειται σε πολύ αυστηρούς όρους. Πρώτον, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε θα δίνουμε τη δυνατότητα εξαίρεσης ε, των ε, παρόχων ε, ακόμη και αν δίνουν τοπικές τιμές. Θα εξακολουθούν να ισχύουν λοιπόν οι τιμές χονδρικής. Μία τέτοιου είδους εξαίρεση από τα διορθωτικά μέτρα θα ήταν ενδιαφέρουσα για τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στις χώρες όπου οι τοπικές τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές. Όμως σε χώρες όπου τα, οι τοπικές τιμές είναι ήδη ανταγωνιστικές και ε, χαμηλές, σε λογικά χαμηλά επίπεδα, προφανώς ε, οι πάροχοι ε, θα θέλουν να εξαιρεθούν γιατί πρέπει να εξακολουθούν να καταβάλουν τις χοντρικές τιμές και ενδεχομένως να έχουν απώλειες αν χρησιμοποιήσουν, αν εφαρμόσουν τις τοπικές τιμές. Υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα με αυτή την προσέγγιση. Δεύτερον, και νομίζω ότι αυτό ετέθη και από κάποιους συναδέλφους σας, ε, η δημιουργία της δυνατότητας ε, εξαίρεσης ή αυτοεξαίρεσης από τα μέτρα ε, αποσύνδεσης, αυτό βέβαια θα αυξήσει το πεδίο εφαρμογής των διαρθρωτικών μέτρων και την δυνατότητα νέων παρόχων να συμμετέχουν στην αγορά Κάτι ε, το οποίο δεν θα ίσχυε αν υπήρχαν, ε, αν υπήρχαν ε, πάροχοι που δεν θέλουν να εξαιρεθούν από τα μέτρα τα διαρθρωτικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αν, λοιπόν, αν υπάρχει αυτή η ρήτρα της αυτοεξαίρεσης να υπόκειται σε πολύ αυστηρούς όρους. Και δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα με, όσους, ε, με τους νέους παρόγους που θέλουν να συμμετέχουν στην αγορά. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ποιος θα εφαρμόσει τη ρήτρα ε, των ε, τοπικών τιμών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε λοιπόν όλε αυτές οι ιδέες, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε επαρκώ. Τώρα ένα μάλλον διαδικαστικό ζήτημα που είναι πώς θα ολοκληρώσουμε τις, τα διαρθρωτικά μέτρα. Υπάρχει επιθυμία, από ό,τι ακούω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει την τεχνική ε, απόφαση για την αποσύνδεση. Ο χρόνος όμως είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον ανταγωνισμό πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο το συντομότερο δυνατόν. Και πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται απαραίτητο να προσφύγουμε σε προηγούμενες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ε, το θέμα αυτό και από ό,τι βλέπω από τι τροπολογίε έχουμε κριτήρια για τα μέτρα αποσύνδεσης και αυτά θα έπρεπε να αποτελούν επαρκή ε, καθοδήγηση για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων. Ε, ο κανονισμός ε, ήδη δίνει αρκετή ασφάλεια δικαίου και εμείς θα μπορούσαμε ίσως να τον συμπληρώσουμε με κάποια μέτρα κατευθυντηρίων γραμμών και στη συνέχεια μπορεί να υπάρξει και μια επιπλέον απόφαση αν τα κατευθυντήρια αυτά μέτρα δεν είναι επαρκή. Αλλά δεν, θεωρούμε, δεν θεωρούμε απαραίτητο να ξεκινήσει μια ακόμη διοικητική διαδικασία ε, γιατί κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο. Και όπως είπα ότι ο, ο χρόνος είναι ε, καθοριστικός παράγοντας εν προκειμένου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν εδώ την παρέμβασή μου και όπως είπα στην αρχή ε, χαιρετίζω τις εργασίες ε, που έχουν λάβει χώρα ως τώρα και ελπίζω να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό κατά τους ερχόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω το λόγο στην κυρία Νίπλερ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όπως είπα και στην αρχή στους συναδέλφους θέλω να τους ευχαριστήσω για τα ενδιαφέροντα σχόλια, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και προσβλέπω και στην περαιτέρω συνεργασία μας. Στρέφομαι προς τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ευχαριστώ για την προθυμία να καταλήξουμε σύντομα σε επικοδομητικές λύσεις προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ζητώ συγγνώμη ε, που οι συμβιβαστικές τροπολογίες δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σύντομα, αλλά αφού σας παρουσίασα τις ε, κεντρικές ε, γραμμές, χαίρομαι ότι βάσει των σχολείων μου μου δώσατε τις απόψεις σας και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Θέλω να απαντήσω σε ορισμένους Συναδέλφου, διότι πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην κατάσταση σχετικά με την περιαγωγή και την ανάλυση του Συμβουλίου. Ο συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά που είπαν επ' αυτού και πιστεύω ότι η συζήτηση έγινε πάρα πολύ επικοδομητικά μπορέσαμε να λύσουμε ορισμένα προβλήματα ε, στην ε, δυστοκία των περιαγωγών και ε, θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τις τροπολογίες σχετικά με το local breakout διότι πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε εδώ επειδή ορισμένοι συνάδελφοι ε, με ρώτησαν ότι το roaming είναι κάτι πεπαλαιωμένο ότι για την παραγωγή πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκές ενιαίες τιμές αυτό είναι σωστό αλλά εδώ είναι αντίθετη η αρχή αυτή στο να υπάρχει ανταγωνισμός και να αφήσουμε την αγορά να διαμορφώσει ε, τις τιμές μόνη της και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι εδώ είμαστε υπέρ του ανοίγματο της της ας αφήσουμε τον σχετικό κλάδο να διαμορφωθεί μόνος του με ορισμένους φραγμούς όσον αφορά τα πλαφόν. Και αυτό θα έχω υπόψη μου και για τη συμβιβαστική λύση, διότι πρέπει να σκεφτούμε μία ενιαία τιμή και αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιθυμούσαμε ε, θα ε, έπρεπε να μην προτείνουμε στις επιχειρήσεις διαρθρωτικά μέτρα. Είτε θα ανοίξουμε την αγορά και θα υποχρεώσουμε τους παρόχους με ε, διαρθρωτικά μέτρα να διευρύνουν την πρόσβαση ή θα τους αφήσουμε να κινηθούν μόνοι τους. Είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτείτε. Ε, σας έχω παρουσιάσει τις εναλλακτικές λύσεις και θα ήθελα να μου πει ποιος είναι υπέρ του ανοίγματο της αγοράς και της ελεύθερης εξέλιξης της αγοράς σχετικά με τα πλαφόν των τιμών. Έχει γίνει συζήτηση όπως ε, αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες. Οπότε μην νομίζετε ότι εδώ το περιθώριο ε, χρειάζεται να διαμορφώνεται για το κέρδος με ε, τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίσει τον ανταγωνισμό αντιθέτως και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους απλώς ε, να θυμούνται ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου εκεί θα γίνει περαιτέρω συζήτηση για τις τιμές ως εκ τούτου ε, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μία λογική πρόταση με την οποία να, ε, ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Όταν, διαβάστε λοιπόν το συμβιβαστικό κείμενο, άπαξε θα το έχετε και όσον αφορά την πρόταση της κυρίας Βάλεαν των φιλελευθέρων θεωρώ ότι η διατύπωση είναι σωστή αλλά επιφυλάσσομαι όταν θα ακούσω τα περαιτέρω σχόλιά σας. Όσον αφορά την ρήτρα opt-out υπάρχουν διάφορες απόψεις. Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή μόνο τρεις χώρες είναι υπέρ του opt-out η Γαλλία, η Ισπανία και η Κύπρος και εγώ έχω εκφράσει τις προσωπικές μου επιφυλάξεις καθότι του ε, ε, ε, οι ελάχιστοι στηρίζουν το opt-out αλλά έχω προτείνει αυτό το συμβιβαστικό θέμα γιατί προσπαθώ σαν τους συναδέλφους να υποκινήσω ένα πιο έντονο ανταγωνισμό και ευχαρίστως να ξανακάνουμε τη συζήτηση όπου τον τελευταίο λόγο θα τον πούμε άπαξ και θα υπάρξει η διερεύνηση της πλειοψηφίας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συμβιβαστικές προτάσεις για να έχουμε ε, χώρο να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση. 15 είναι οι ε, ε, συμβιβασικέ τροπολογίες και αν θέλετε στην επόμενη συνεδρίαση θα είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε παρατηρήσεις διότι θα δούμε κατόπιν αυτού πόσο θα προχωρήσει αυτό κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην ε, ψηφοφορία ε, με μία ενιαία βάση και να πάμε συσπηρωμένοι στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, όπως είπα, να, να έρθετε σε επαφή μαζί μου για τις συμβιβαστικές προτάσεις εάν κάτι ακόμη σας ενοχλεί. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία στις επόμενες εβδομάδες για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Εάν κάποιος άλλος δεν θέλει να λάβει τον λόγο, τότε εγώ θα ήθελα ήθελα να σταματήσω αυτή τη συνεδρίαση η οποία θα ξαναξεκινήσει σε 20 λεπτά με τον, τη συνάντηση με τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό, τον κύριο Μάρτιν Λίντεγκαρντ για τα, το κλίμα, την ενέργεια και τις κατασκευές. Ευχαριστώ.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 μόνο Bene, allora... Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας ε, τον Δανό Υπουργό για το κλίμα, την ενέργεια και τις κατασκευές, ο οποίος ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον ε, κύριο Μάρτιν Λίντεγκαρντ. Τον καλωσορίζουμε εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής. Ε, έχουμε στη διαθεσή μας τρία τέταρτα για την συνάντηση αυτή και κατόπιν ε, θα έχουμε ε, μια δεύτερη επίσκεψη από έναν άλλον Υπουργό. Θα ακούσουμε λοιπόν καταρχάς τον Υπουργό, κατόπιν έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα για τρία λεπτά, απάντηση από τον Υπουργό και κατόπιν θα λάβουν το λόγο οι υπόλοιποι Ευρωβουλευτές. Το λόγο έχει ο Υπουργός Λίντεγκαρτ, τον οποίο καλωσορίζουμε και πάλι εξ ονόματος όλων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας. Θα ήθελα καταρχάς κύριε Πρόεδρε να σας, να σας συγχαρώ για το ε, διορισμό σας ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω ε, στην Επιτροπή σας ε, τι προτεραιότητε τη Δανική Προεδρίας. Όπως γνωρίζετε έχουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα ε, μπροστά μα και θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα τα οποία θα καλύψουμε. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει, να τα καλύψω σχεδόν όλα γιατί πρέπει να αποφασίσουμε το μέλλον του τομέα της βιομηχανίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τους επόμενους έξι μήνες. Όπως γνωρίζετε, ε, βασική ανησυχία των κρατών μελών και των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα έπρεπε να είναι η κατάσταση των, ε, της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ε, των χρηματοοικονομικών και οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα έπρεπε να ε, ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, να αυξήσουμε την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και να ε, θωρακίσουμε τις οικονομίες μας από τιμολογικές διακυμάνσεις λόγω των ενεργειακών τιμών. Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφή πολιτική. Πρέπει να έχουμε σαφή ορόσημα για την ανάπτυξη ε, της ενέργειας ε, και της πολιτικής για το κλίμα ε, μέχρι το 2030-2040. Επίσης πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και να επιτύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2020. Γι' αυτό ακριβώς εμείς έχουμε έναν από τους τέσσερις πυλώνες της Δανικής Προεδρίας, την Πράσινη Ευρώπη. Όχι, όχι παρά την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως λόγω αυτής. Έχουμε θέσει το στόχο της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης ε, κατά 20% μέχρι το 2020, το να χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά την ενέργεια δηλαδή. Ο λογαριασμός του πετρελαίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 ήταν 315 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση πάνω από 40% σε σχέση με το 2020, δηλαδή κάτι παραπάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ και λόγω των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου κυρίως. Πρέπει λοιπόν η ανάπτυξή μας να καταστεί πιο πράσινη, να διοχετεύσουμε ε, κονδύλια στις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να μεταφέρουμε τις επενδύσεις μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα βασικός τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι η συμφωνία επί της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ε, και να εξοικονομήσει ενέργεια, αλλά και μπορεί να εξοικονομήσει τεράστια ε, ποσά από, τις, από, τις, από την εισαγόμενη ενέργεια. Μπορεί να είναι μάλιστα ε, ένας τρόπος οικονομικής ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι μπορεί έτσι να δημιουργηθούν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, κάποιες από τις οποίες δεν μπορούν να αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. Κάποιοι μπορεί να ανησυχούν ε, για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί καταλαβαίνω ότι οι ανησυχίες είναι διαφορετικές μεταξύ των κρατών μελών, αλλά στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο η σχέση κόστους αποτελέσματος είναι βασική προϋπόθεση για, την, ε, για την, ε, τον καθορισμό πολιτικών. Και Γι' αυτό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τους, τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει το κενό του 20% να καλυφθεί. Τα μέτρα λογικά θα έπρεπε να επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου αυτού και πρέπει τα μέτρα να αντικατοπτρίζουν ε, τις ε, εθνικές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ε, ευέλικτοι όσον αφορά τα μέτρα. Η έγκαιρη έγκριση ενό τέτοιου νομοθετήματο είναι βασική προτεραιότητα τη Δανική Προεδρία. Ε, Χαιρετίζουμε λοιπόν την εργασία του κ. Τούρμε, που είναι ο εισηγητή, και ελπίζω ότι θα ε, βρούμε κοινό έδαφο μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Φτάνω τώρα στον Ενεργειακό Οδικό Χάρτη 2050 και τον Οδικό Χάρτη για την Οικονομία Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Άνθρακα μέχρι το 2050. Έχουμε Πρέπει να ανανεώσουμε τις ε, συζητήσεις ε, και για τους δύο οδικούς χάρτες ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και ελπίζω να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς αυτό το Μάρτιο. Θέλουμε να εστιάσουμε τις διαπραγματεύσεις για την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ενεργειακό Οδικό Χάρτη για το 2050 ε, γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη βάση για μακροπρόθεσμες αποφάσεις ε, που δίνουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης από τον άνθρακα, ε, ασφάλειας ανεφοδιασμού και ανταγωνιστικότητας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η χρήση ενεώσιμων πηγών ενέργειας είναι στο επίκεντρο των σεναρίων του ενεργειακού οδικού χάρτη. Εκτός από τους δύο δικούς χάρτες, πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή η απόφαση αυτή ε, για το 2030 και 2040 μπορεί να βοηθήσει ε, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές και ε, Γι' αυτό το λόγο ε, είμαι διατεθειμένος να συζητήσω πολύ συγκεκριμένα βήματα για το πώς θα έχουμε ένα ενεργειακό τομέα με λιγότερο άνθρακα. Ε, στις 7 Φεβρουαρίου θα γίνει μια ε, υψηλού επίπεδου διάσκεψη των εμπλεκομένων φορέων εδώ στις Βρυξέλλες και ελπίζω να σας συναντήσω εκεί. Επίσης, ε, η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών δικτύων είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί αυξάνει τα αποθέματα φυσικού αερίου, τις προμήθειες φυσικού αερίου, και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζουμε να έχουμε ε, τη σωστή υποδομή ώστε όλα αυτά να γίνουν με λογικό κόστος. Χρειάζονται επενδύσεις, ε, ε, είναι ένας τρόπος πριμ που μπορούμε να πληρώσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις έτσι ε, από τη μία πλευρά έχουμε αυξανόμενη ζήτηση, χαμηλότερα αποθέματα, τα μεταβλητότητα των τιμών και από την άλλη έχουμε την ανάγκη αντιμετώπισης αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας ε, στα δίκτυά μας ε, και, και την ανάγκη μεταφοράς της ενέργειας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ έγκαιρη. Εγώ δεσμεύομαι να προσπαθήσω να σημειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερη πρόοδος, ε, όμως ε, το θέμα της χρηματοδότησης ε, θα, θα αποφασιστεί τελικά από τους Υπουργούς Οικονομικών. Είναι σε πρώιμο στάδιο ακόμα και η όλη διαδικασία και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και τη δουλειά του κυρίου Κορέα Ντεκάμπος προς αυτό. Επίσης, ε, η έκθεση ιδίας ε, πρωτοβουλίας κυρίας Χέρζοκ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Ε, όσον αφορά τώρα τις διακυβερνητικές συμφωνίες ε, για το αέριο, θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, ε, διαφάνεια και την συνοχή σε εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα... Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να ζητούν σεβασμό των κανόνων της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο διαπραγματεύεται μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με ε, σκοπό να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού, ο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο κύριος Καρίνς. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε μαζί του με ε, συμβιβαστικό πνεύμα. Υπάρχουν σημαντικέ διαφορές και κατακαιρματισμό μεταξύ των ε, νομοθεσιών των κρατών μελών, αλλά και των πρακτικό του. Ε, μετά τι συνέπειες τη καταστροφή ε, στο κόλπο του Μεξικού το 2010, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειώσουμε τέτοιου είδους κινδύνου στα ευρωπαϊκά ύδατα. Ε, αν υπάρξει τέτοιου είδους καταστροφή. Ε, θέλουμε λοιπόν να αφιερώσουμε ε, πολύ χρόνο στις offshore δραστηριότητες εξόριξης πετρελαίου και αερίου. Και Όσον αφορά τώρα την, το σήμα Energy Star, η, Ευρωπαϊκή, η Προεδρία της Δανίας θα προσπαθήσει να ε, εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία με το ε, Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και αναμένω εναγωνίω την συνεργασία και τις συζητήσεις μας κατά τους επερχόμενους έξι μήνες. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση τώρα. Η κυρία Ντελκαστίγιο για τέσσερα λεπτά. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό για την σημερινή του παρουσία εδώ. Να πω καταρχάς τον Δανό Υπουργό, όπως έλεγα και στο Δανό εχθές Υπουργό που ήρθε για την ενέργεια εδώ να συζητήσουμε για το ορίζον 2020, ότι βρίσκεστε σε μία αξιοζήλευτη θέση ως Προεδρία. Πραγματικά ε, σας φθονούν οι υπόλοιπε Προεδρίες γιατί έχετε δύο ζητήματα τα οποία ε, είναι πρώτου μεγέθους πραγματικά. Το ένα είναι ενεργειακή απόδοση η οποία προχωρά και ε, το άλλο είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα που είναι το μεγάλο πρόγραμμα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα από τα προγράμματα που έχουν το μεγαλύτερο κοινοτικό προϋπολογισμό. Επομένως, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να σας συγχαρούμε που βρίσκεστε ε, στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όταν συζητώνται τα θέματα αυτά θα έχουμε καλή συνεργασία ελπίζω. Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση υπάρχει πολύ μεγάλη συνένεση ως προς το πιο ουσιώδες ζήτημα. Συμφωνούμε όλοι ότι απαιτείται αποτελεσματική κατανάλωση της ενέργειας για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, για λόγους μείωσης των εκπομπών και τρίτον, για ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά νέο, αλλά το οποίο αυξάνεται συνεχώς, που είναι το οικονομικό πρόβλημα, σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά οικονομική κρίση που βιώνουμε και η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα καλό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης, ένα καλό σχέδιο ενεργειακής απόδοσης. Εκεί που έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα είναι το πώς. Οι στόχοι είναι σαφείς και η σημασία τους είναι σαφείς. Το πώς είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και υπό αυτήν την έννοια υπάρχουν δύο πτυχές οι οποίες θα ήθελα να επισημάνω και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τις συζητήσουμε και αλλού. Καταρχάς, η έννοια της ενεργειακής απόδοσης υπό την έννοια της ενεργειακής αποταμίευσης απλώς και μόνο και εγώ θεωρώ ότι ε, θα ε, εκφράζω και την άποψη της πολιτικής μου ομάδας εδώ ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της ενεργειακής έντασης όταν αναφερόμαστε στον κλάδο διότι δάλλως δεν θα μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη ή κατά κάποιο τρόπο θα εξαντλούμε τις δυνατότητες ε, οικονομικής ανάπαξης. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στον κλάδο, η έννοια της ενεργειακής έντασης και η εφαρμογή της έχει μεγάλη σημασία και ένα δεύτερο το οποίο μου φαίνεται ζωτική σημασία κύριε Υπουργέ είναι τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, είναι ε, πολύ διαφορετική από πλευράς κλίμακος, ε, δημογραφικού ε, και σε οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από αυτούς που διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή τα κράτη-μέλη, που να μπορούν να αναπτύξουν ένα σύνολο μέτρων τα οποία θα είναι ισοδύναμα ως προς τα αποτελέσματα που προτείνονται, θα έχουν ταυτόχρονα και τη δέουσα ευελιξία. Η έννοια της ευελιξίας είναι θεμελιώδης διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά δεν υπάρχει καλύτερος κανόνες από αυτός που εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Το να έχουμε ένα κανόνα ο οποίος ε, κατά την εφαρμογή του, κατά την εξέλιξή του δεν προσαρμόζεται όπως ε, πολλές φορές συμβαίνει σε αυτό που λέει η οδηγία δεν μας ε, χρειάζεται για τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια δέσμευση ώστε να υπάρχει ευελιξία η οποία θα μας οδηγήσει στα ισοδύναμα αποτελέσματα ε, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό για την πολιτική μας ομάδα είναι ζωτική σημασία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε επισταμένα με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Τόμψον. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Για μας είναι μεγάλη χαρά και ε, θέλαμε να μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο με τον ε, Υπουργό που είναι αρμόδιος ε, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και να μπορέσουμε να συζητήσουμε την σχετική οδηγία αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν συζητήσαμε το θέμα της χρηματοδοτήσεως. Τι εννοώ με αυτό. Βλέπουμε ότι οι εξοικονομήσεις ενεργείας σε όλους τους τομείς, είτε μιλάμε για την βιομηχανία είτε για τα κτίρια, είναι θέματα σημαντικά για την εξοικονόμηση ενεργείας αλλά χρειάζονται πολλά χρόνια μέχρι ότου να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την εξοικονόμηση και χρειάζονται μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είναι λοιπόν αναγκαίο κατά τη γνώμη μου να διατεθούν ορισμένοι πόροι στα νέα κράτη-μέλη διότι πολλά νέα κράτη-μέλη φοβούνται ότι αυτή η οδηγία για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα είναι πολύ δαπανηρή και αναρωτιέμαι πώς εσείς σκοπεύετε να διαχειριστείτε ε, τα διαρθρωτικά ταμεία και ε, να τα χρησιμοποιήσετε για χρηματοδότηση διότι είχαμε πει προετών να εξοικονομήσουμε ορισμένα κονδύλια από τα ε, διαρθρωτικά ταμεία για την χρηματοδότηση της ενεργείας και τώρα τα εθνικά κοινοβούλια μας έχουν παρακαλέσει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο ποσό για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στον προϋπολογισμό των διαρθρωτικών ταμείων διότι διαφορετικά δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος διότι όλοι θα προτιμήσουν νέους αυτοκινητοδρόμους παρά εξοικονόμηση ενεργείας Πρέπει λοιπόν να δούμε αν ε, το Περιφερειακό Ταμείο μπορεί να ε, καθορίσει συγκεκριμένα κονδύλια για την αποτελεσματικότητα της ενεργείας, αν αυτό θα μπορέσει να συνάδει με τη δημιουργία 2 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, τις οποίες ε, έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι χρειαζόμαστε για τις αυτές Συγκεκριμένε συγκεκριμένες ε, δεξιότητες και ε, εμπειρούς τεχνικούς. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω στην αρμόδια επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε για να ε, έχουμε κοινούς στόχους χρηματοδότησης που μου φαίνονται πολύ σημαντικοί. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς θα καταλήξετε σε αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζω τα σχόλια τα οποία έγιναν σχετικά με ε, τις ε, επόμενες κινήσεις. Καταρχήν ήθελα να αναφέρω ότι το σημείο κίνησης των διαφορετικών κρατών μελών είναι ε, διαφορετικό αυτή τη στιγμή και έτσι για την ε, οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητας ε, υπάρχουν διαφορετικές αξιολογήσεις και ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, όπως συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτικούς ήδη στόχους στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και ανησυχούμε διότι η ε, εξέλιξη ε, στο Συμβούλιο στο θέμα των δεσμευτικών στόχων δεν έχει προχωρήσει όπως θα επιθυμούσαμε. Μπορείτε εσείς να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η κατάσταση στο Συμβούλιο εάν δηλαδή έχει υπάρξει μία αλλαγή στη θέση των κρατών μελών σχετικά με τους δεσμευτικούς στόχους ή αν υπάρχει ακόμη μία μεγάλη πλειοψηφία η οποία είναι είναι αντίθετη. Επίσης χαιρετίζω το γεγονός ότι έχετε τονίσει τη σημασία του κλίματος διότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εισάγουμε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου και πληρώνουμε τιμήματα τα οποία δεν μπορούμε να ανθέξουμε. Ίσως λοιπόν θα πρέπει βάσει των συζητήσεων που έχουν γίνει στο Συμβούλιο να υπάρξει μία ανάλογη κίνηση όπως αυτή της εξέτασης της ενεργειακής αποτελεσματικότητος δηλαδή να υπάρξουν ορισμένες υποχρεώσεις που θα επιβληθούν στις δημόσιες αρχές διότι ε, αυτές ε, ε, ε, αυτός είναι ο χώρος όπου εμποδίζουν την εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου άρθρου και θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και ποιο είναι το κείμενο της οδηγίας το οποίο θα μπορούσε να είναι εφικτό. Ξεκινώντας από την κυρία Ντεκαστήγιο τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι αντιλαμβάνουμε ότι μέχρι στιγμής έχει υπάρξει σύγχυση. Ορισμένοι θεωρούν ότι η ενεργειακή οδηγία θα οδηγήσει σε μία μείωση κατά 80% σε σχέση με το 2007 παρόλο που ορισμένοι θα ήταν ευχαριστημένοι αλλά ε, ε, η Επιτροπή λέγει ότι θα υπάρξει μείωση 80% αν το συγκρίνουμε με ανάπτυξη και αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε προς τα που κατευθυνόμαστε και εάν απλώς θα υπάρχει ένας στόχος απλώς έντονης προσπαθίας ο οποίος ίσως προχωρήσει την κατάσταση βράχη πρόθεσμα αλλά δεν θα οδηγήσει σε μια πραγματική οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη. Ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ όταν όλες τις τιμές ανεβαίνουν, τα περισσότερα, οι περισσότερες συμφωνίες αερίου που ε, παρέχουν αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έναν τιμάριθμο. Ε, πέρσι έχασαν τεράστια, ε, χάθηκαν τεράστια ποσά γιατί τα, οι τιμές που προβλέπουν οι συμφωνίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Πρέπει λοιπόν να εξαρτώμαστε λιγότερο από τις εισαγωγές αυτές. Διαφορετικά τα οικονομικά μας και η γεωπολιτική μας ε, θα ε, απειλούνται, να μην πω ότι θα είναι αντικείμενο εκβιασμού. Υπάρχει ένα ε, βασικό ζήτημα, η ένταση της ενέργειας. Έχω δίκιο όταν λέω ότι αν η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία και όλες οι υπόλοιπες χώρες που έχουν αρνητικό ΑΕΠ αν έχουν ένα στόχο ενεργειακής έντασης. Αυτό θα σήμαινε, κατά τη γνώμη μου, ότι θα ήταν αδύνατο για τις χώρες αυτές να επιτύχουν έναν τέτοιο στόχο. Έχουμε κάνει κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς ότι ακόμη για την Πολωνία που είχε το τέταρτο, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, ότι ένας στόχος ενεργειακής έντασης ε, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί για να ε, δεν θα μπορούσε να το αντέξει ε, η συνολική οικονομία. Γι' αυτό στο κείμενο του Συμβουλίου οι κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ επιφυλακτικές για την αναφορά ε, της ενεργειακής έντασης ε, ως δείκτη. Ε, πώς καταφέρατε εσείς στη Δανία να υπερβείτε αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας και της πολιτικής ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας που είναι υποχρέωση στην Δανία, πώς επηρεάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα ώστε να ε, προκαλέσει ε, επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα στη Δανία. Και ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο το ανέφερε και η κυρία Τόμσεν είναι η χρηματοδότηση. Το γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επειδή υπήρχε κίνδυνο να χάσει το τριπλό α, μείωσε ριζικά ε, τα δραστικά τα ε, ε, δάνεια, τα δάνειά της. 67 δισεκατομμύρια ε, επενδύσεων γίνονταν στην ευρωπαϊκή οικονομία ε, και μάλιστα σε ευρωπαϊκά προγράμματα μηγός έχουν αποφασίσει από τα 67 να πέσουν στα 50 δισεκατομμύρια και αυτό είναι λόγω των οργανισμών ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης επειδή φοβούνται μη τυχόν τους υποβαθμίσουν. Υπόθηκε, έμαθα λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων μπορεί να υπάρχει σημαντική πολιτική συμφωνία που θα ήταν η εξή. Ε, τα υπόλοιπα των διαρθρωτικών κειμένων, ε, των διαρθρωτικών ταμείων, ε, πολλά δισεκατομμύρια, να τα μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα δώσει τη δυνατότητα να, δώσει τη δυνατότητα να αυξήσει πάλι τα δάνεια που δίνει δεν μπορώ να, δω, να σκεφτώ τίποτα άλλο που θα μπορούσε να προκαλέσει επενδύσει στην πραγματική οικονομία και στα πραγματικά προγράμματα υποδομών από αυτό το μέτρο που μόλι σας ανέφερα. Επειδή λοιπόν εσεί βρίσκεστε στη θέση του οδηγού και επειδή ο Πρωθυπουργό σα θα πάει στο Συμβούλιο που ανέφερα το, τη Δευτέρα, ποια είναι η θέση λοιπόν τη Δανίας όσον αφορά το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όταν, μιλά, όταν μιλάμε για, ε, πραγματικές, ε, για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, οικονομία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δώσουμε το λόγο στον Υπουργό τώρα για να απαντήσει σε αυτό τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τις πολιτικές ομάδες και μετά θα έχουμε τις ερωτήσεις από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα πολύ εύστοχα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με την κυρία Πιλάρ Τελκαστήγιο. Και αυτό εν μέρη θα πατά και στην κυρία Χολ για τους δεσμευτικούς στόχους και τους εντατικούς στόχους. Για να είμαι ειλικρινής, ε, χρειάστηκε να συζητήσουμε τους δεσμευτικούς στόχους πριν από κάποια χρόνια στο Συμβούλιο, αν θυμάστε καλά, και δεν βλέπω κάποια αλλαγή ε, στη θέση των κρατών μελών. Τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο μέχρι τούδε. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο, κατά πάσα πιθανότητα, θα εμείνουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε δεσμευτικά μέτρα. Και αυτό εν μέρει απαντά και στον κύριο Τούρμες. Νομίζω ότι η παρούσα απόφαση είναι ότι θα εμείνουμε στα δεσμευτικά μέτρα και κάποια θα λάβουν υπόψη τους και το ποσοστό ανάπτυξης και από εκεί και πέρα το 2014 και 2015 θα αξιολογήσουμε πώς προχωρούν τα πράγματα και ε, θα δούμε αν κινούμαστε προς τον κοινό στόχο και μπορεί να ε, επανεξετάσουμε το ζήτημα για να δούμε αν χρειαζόμαστε κάτι επιπλέον. Για να το επιτύχω, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ ακριβέ αριθμητικό στοιχείο, γι' αυτό και ακριβώ και σε αυτό εμένουμε στην πρώτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Φιώνα Χολ που λέει ότι στο στόχο που έχουμε επί του παρόντος έχουμε συμπεριλάβει και ένα ποσοστό ανάπτυξης και νομίζω ότι ε, το Συμβούλιο πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στα μέτρα. Και εδώ συμφωνώ απολύτω και νομίζω ότι το Συμβούλιο συμφωνεί απολύτω ότι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη ελαστικότητα, διότι η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Εκεί που δεν μπορούμε να είμαστε ελαστικοί στο είναι στο γεγονό ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Και αυτή είναι η θέση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν υπάρχουμε ευελιξία στα μέτρα θα πρέπει όλα τα μέτρα να έχουν ως στόχο την επίτευξη του κοινού αντικειμενικού σκοπού. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στη διαδικασία πρέπει πράγματι να πούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας για να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν ε, με διάφορους τρόπους στην κάθε χώρα ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος το συντομότερο δυνατόν. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Δημιουργήθηκε μια παρέμβαση λόγω των ακουστικών. Τώρα, η κυρία Τόμψεν και ο κύριος Τούρμεν αναφέρθηκε στο θέμα της χρηματοδότησης και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε μικρή κλίμακα ε, χρηματοδότηση, χρηματοδότηση των κυριών για παράδειγμα, αυτά τα έχουμε στην παρούσα πρόταση. Υπάρχει κάποια πρόταση μικροχρηματοδότησης. Αν δείτε για παράδειγμα την πρόταση για το δημόσιο και για τις επιχειρήσεις, αλλά όταν φτάνουμε στα πιο στρατηγικά, στα πιο μεγάλα ζητήματα χρηματοδότησης, ίσως καλό θα ήταν με την προσέγγιση μέσω διαρθρωτικών ταμείων και διάφορων άλλων στρατηγικών θεμάτων που θα λάβουμε υπόψη. Όπως σας είπα όμως, ε, και στην αρχική μου παρέμβαση ότι δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Αυτή είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία για τα κράτη-μέλη, για το ΕΚΟΦΗΝ και για την αρχή προπολογισμού. Εγώ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσω λοιπόν να προχωρήσω περαιτέρω στο θέμα αυτό, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα ε, πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση σίγουρα δεν θα επιτύχουμε τους κοινού μας στόχους. Για την ερώτηση για το δημόσιο τομέα που έθεσε η κυρία Φιώνα Χόλ. Η αίσθησή μου είναι ότι όσον αφορά το δημόσιο τομέα, ε, ο, και τι μπορούμε να θέσουμε ως απέτηση στους Δήμους, πολλά κράτη-μέλη ε, ρωτούν τι μπορούμε να κάνουμε προς αυτό το τομέα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας όμως ότι ε, Τη όλη διαδικασία πρέπει να ηγηθεί ο δημόσιο τομέα. ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο τμήμα του δημόσιου τομέα τελικώς θα έχουμε στην τελική συμφωνία. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Τούρμε για την περίπτωση της Δανίας, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πριν από τέσσερα χρόνια ε, ξεκινήσαμε την αγορά για την ενεργειακή εξοικονόμηση και όπω πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εταιρείε ενέργεια χρειάστηκε να ανταγωνιστούν για να δούνε τι χρειάστηκε να κάνουν. Μπορούσαν να έχουν ένα όφελο, αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να βοηθήσουν του καταναλωτέ να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργεια. Και τότε και ο κλάδο και οι επιχειρήσει ενέργεια ήταν κατά τη διαδικασία γιατί θεωρούσαν ότι θα ήταν πολύ δαπανηρή. Το θέμα είναι ότι σήμερα ξαναγίνεται αυτή η συζήτηση και τώρα και οι ενεργειακές επιχειρήσεις και ε, ο κλάδος είναι στο γραφείο μου και μας πιέζουν να αυξήσουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης για να διευρύνουμε την αγορά, διότι από ό,τι φαίνεται ε, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά ε, χρήματα και μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ περισσότερα χρήματα μέσω αυτού του ανταγωνισμού ε, και έτσι εξοικονομούν ενέργεια. Και έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας με πολύ φθηνό τρόπο. Ε, σας ζητώ λοιπόν να ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα διότι μας εξέπλεξαν τα αποτελέσματα και το να συμμετέχει ο ίδιος ο κλάδος, η αγορά, ε, να υπάρχει ανταγωνισμός ε, όπου θα είναι κινητήριος μοχλός όλης αυτής της εξέλιξης σίγουρα θα είναι προς όφελός μας. Τώρα, νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε 7 εγγεγραμμένους στον κατάλογο για 6 λεπτά και θα κλέψουμε ένα-δυο λεπτά για να δώσουμε απαντήσεις. Ένα λεπτό ο καθένας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Κύριος Μπαλσίτη. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως η Ιδανική Προεδρία είναι πάρα πολύ ε, φιλόδοξη και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν οπότε ε, θα πρέπει όμως για πολλά να περιμένουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι αποφάσεις αυτές δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν εύκολα. Πράγμα το οποίο σημαίνει όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα ότι ε, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και ορισμένες φορές απογοητευόμαστε ή προσπαθούμε να αποκρύψουμε την πραγματικότητα ημένα από τους δε. Και εδώ αναφέρουμε στη δημιουργία των υποδομών, τις οποίες χαιρετίζω, αλλά σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς σχετικά με τους μηχανισμούς τιμών διότι ξέρουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν χρειάζεται δεν δημιουργεί επιπρόσθετες ε, επιβαρύσεις από πλευράς κόστος υπάρχει ε, ένας ε, ε, ηλεκτρικός σταθμός. Εάν λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τιμές και τους μηχανισμούς των τιμών και εδώ αναφέρομαι στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις ε, ε, διαπραγματεύσεις για την αγορά ε, πρώτων υλών δημιουργίας ενεργείας από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχω μία ερώτηση προς τον Υπουργό σχετικά με την οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητος, διότι συνήθως δεν είμαστε υπέρ των δεσμευτικών μέτρων αλλά υπάρχουν τα δεσμευτικά μέτρα και θέλει να επιμείνει σε αυτά και ο Υπουργός. Πώς φαντάζεται λοιπόν ότι θα μπορέσει να τα επιβάλλει διότι όταν λέει ότι το, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και πολλοί στο Κοινοβούλιο είναι πεπισμένοι ότι δεν πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικά μέτρα θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και το θέμα της ε, αποδομήσεως των σταθμών. Πρέπει παρόλα αυτά να, να διατηρήσουν τις επενδύσεις στις βιώσιμες ενέργειες. Οπότε εσείς ε, πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να προωθήσετε τα θέματα αυτά για να καταλήξετε μια συμφωνία σχετικά με την ενεργειακή ε, ασφάλεια. Ε, ο κύριος Μπούζεκ, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που επανέρχομαι στην Επιτροπή Ήτρε μετά από δυόμιση χρόνια. Εχθές ήμουν στην Επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων αλλά σήμερα εδώ αισθάνομαι σπίτι μου και χαίρομαι που βλέπω τόσους συναδέλφους γύρω μας. Μία πολύ σύντομη ερώτηση και ίσως καλύτερα να την εκφράσω στη γλώσσα μου, τα πολωνικά. Ε, Έχουμε μεγάλες ε, ελπίδες από την ε, Δανική Προεδρία σχετικά ε, με την επιβολή του κλιματικού πακέτου. Είστε οι πρωταθλητές της Ευρώπης, έχετε τις καλύτερες λύσεις και παράγετε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρησιμοποιεί η χώρα σας σχετικά με μία ανάλυση κόστους για να μπορέσει κανείς να κατανείμει το κόστος αυτό αναχώρες. Ακούσαμε ότι ορισμένα κράτη έχουν πρόβλημα για να εφαρμόσουν ορισμένους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αυτή τη στιγμή εξετάζει το θέμα και χρειάζεται μία ανάλυση του κόστους και της κατανομής αναχώρα ε, στην ευρωπαϊκή αγορά για να μπορέσουμε ε, να εστιαστούμε στο σωστό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δανική Προεδρία για την παρουσία της, ε, να της ευχηθώ κάθε επιτυχία για τους επόμενους έξι μήνες. Έχω μία ερώτηση για το, για το ε, πρόγραμμα Horizon 2020. Ε, οι καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες ε, είναι ένα σημαντικό τμήμα του, της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 16 δισεκατομμύρια για την κλιματική μεταβολή και τις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες. Έχουμε λοιπόν τις σωστές προτεραιότητες, έχουμε τις σωστές επιλογές, προκειμένου η αηφορία να μπορεί να συμβαδίσει με την ανταγωνιστικότητα και χαίρομαι που είδα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα στο, στη βιομηχανία έχει επανέλθει ως προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τις σωστές προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε όμως και τα σωστά μέσα, γιατί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είχε επικεντρωθεί πάρα πολύ στην έρευνα. Η ενέργεια χρειάζεται επίσης ε, πάρα πολλά προγράμματα ε, επίδειξης για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν τα ενεργειακά προγράμματα. Και έχω και μία ερώτηση όσον αφορά την εξερεύνηση για τα αποθέματα ε, όπως επίσης και για την πρόληψη των ατυχημάτων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων στο Συμβούλιο γιατί κάποιες χώρες έχουν ήδη νομοθεσία αλλά η κατάσταση διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα κινηθεί η ε, Δανική Προεδρία σε σχέση με αυτό. Panie ministrze, powiedział pan, że jednym Ένας από τους δεσμευτικούς στόχους είναι η μείωση ε, της ενέργειας κατά 20%. Επίσης, θέλουμε να μειώσουμε την αποτελεσματικότητα κατά 20%, να αυξήσουμε συγγνώμη, την αποτελεσματικότητα κατά 20%. Αλλά αυτός είναι ο συνολικός στόχος και όχι ο στόχος αναχώρα, διότι θα πρέπει να το υπολογίσετε σε ΑΕΠ κατά κεφαλήν ε, ε, για την κάθε χώρα. Ε, χρησιμοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία και τη Eurostat το 97 ως χρονιά αναφοράς για να φτάσουμε μέχρι το 2020. Εγώ θα ήθελα να ξέρω με ποιο τρόπο υπολογίζεται την ενεργειακή απόδοση. Η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ η Ιδανική Προεδρία έρχεται σε συνέχεια της Πολωνικής Προεδρίας και συνεργαστήκαμε σε πολλά ζητήματα και αυτή τη στιγμή είναι πλέον η σειρά σας να αναλάβατε κάποια θέματα και κάποια προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας. Όπως για παράδειγμα η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι οι διακυβερνητικές συμφωνίες σε θέματα ενέργειας. Και η ερώτησή μου είναι εξής. Στο έγγραφο για τις διακυβερνητικές συμφωνίες αναφέρεται ότι κάποιες από τις συμφωνίες θα είναι εμπορικής φύσεως, ενώ κάποιες άλλες θα καλύπτονται από τις διακυβερνητικές συμφωνίες. Στις διακυβερνητικές συμφωνίες θα γίνεται έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αν είναι καθαρά εμπορικής φύσεως οι συμφωνίες, από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις ε, ε, ε, διαπραγματεύσεις. Το πρόβλημα είναι πώς θα καθορίσουμε ποιες συμφωνίε είναι αυστηρά εμπορική φύσεως και κάποιες άλλες είναι διακυβερνητικές ε, για άλλα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι εγώ θεωρώ και έχω καταθέσει και σχετική τροπολογία και κάναμε και σχετική συζήτηση επί του ζητήματος αυτού εχθές εδώ στην Επιτροπή μας Θεωρώ λοιπόν ότι και για τις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει έλεγχο ώστε οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να παίζουν με τους ορισμούς διότι μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται εμπορική συμφωνία αλλά δεν θα γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος και δεν θα το γνωρίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ σαφείς προς τους ορισμούς. Είχαμε ξεχάσει τον κύριο ε, Ρομπ ω τελευταία παρέμβαση. Έχουμε ξεφύγει λίγο από τα χρονικά όρια. Θα αφήσουμε τρία λεπτά στον Υπουργό για να απαντήσει. Μία ερώτηση λοιπόν μόνο προ τον ε, Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι, κύριε Υπουργέ. Να ρωτήσω λοιπόν τον Υπουργό κατά πόσον γνωρίζει ότι στην πρόταση για τις υποδομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο αποθεματικό για την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα λοιπόν για τα ευρυζωνικά δίκτυα από τις υποδομές ενέργειας. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον σκοπεύετε να ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό, διότι αν θέλετε να κάνετε κάτι για την πράσινη ενέργεια στο μέλλον και ελπίζω να συμφωνούμε όλοι ότι μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για να μεταφέρεται η ενέργεια. Και ε, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ευρώπη στο ζήτημα αυτό. Ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Τώρα θα προσπαθήσω να σας απαντήσω χωρίς να έχω πάρα πολύ χρόνο οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα αλλά είχαμε πολλά θέματα που συζητήσαν. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλα αυτά είναι διότι ε, ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι, ξέρουμε τις ε, τι τις οποίες κάνουμε για δεσμευτικούς στόχους αλλά ε, ε, ε, στο Συμβούλιο αυτό ακριβώς συζητάμε. Δεν βλέπω να υπάρχει αλλαγή. Δεν ξέρω αν στο μέλλον θα υπάρχει μια αλλαγή πορείας του Συμβουλίου αλλά πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε είναι να υπολογίζουμε τους στόχους και να δούμε πώς ε, θα συμπεριλάβουμε τους σωστούς αριθμούς ε, στην εξέταση αυτή. Ε, σχετικά με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπούσεκ. Βεβαίως, πολύ σωστά είπε ότι κάθε κράτος κοιτάζει ε, το βασικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα το έχουμε προσυζήτηση στη συνάντηση του Μαρτίου όπου ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε, ορισμένες, ε, σε ορισμένα συμπεράσματα. Μετά, σχετικά με, το χρήσιμο ορισμένων εγκαταστάσεων, το οποίο συζητήθηκε και εχθές και ε, ιδίω με τις πολύ χαμηλές ε, τιμές οι οποίες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από όταν ε, είχαμε ξεκινήσει ε, να, εξετάζουμε αυτό το σύστημα. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουμε είναι να αναμορφώσουμε το χρονοδιάγραμμα για το 2030 για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την επιζήτηση των στόχων μας. Το εάν αυτό θα επιτευχθεί είναι κάτι που πρέπει να δούμε διότι εμείς προσπαθούμε να δούμε εάν μπορούμε στον τριμερή διάλογο να καταλήξουμε κάπου και αν έχουμε αριθμούς οι οποίοι είναι λογικοί θα δούμε εάν αξίζει να κλείσουν ορισμένες εγκαταστάσεις. Η κυρία Κουλάσχα Μπαμπίνσκα σχετικά με το IGA. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για να το προωθήσουμε στο Κοινοβούλιο. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε τη συνθήκη και ε, τις, ε, τα συμπεφωνημένα. Πρέπει δηλαδή να λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των κρατών μελών. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διακυβερνητική συνθήκη. Ο κύριος Μπαλκίτης τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και ιδίως ε, για ό,τι είπατε για την υποδομή. Ε, όντως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία καλή τιμή και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα λάβουμε υπόψη μας ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε εξ ονόματος όλων τον Υπουργό για αυτή την πρώτη του παρουσία εδώ. Είμαι βέβαιη ότι θα το ξαναδούμε επανειλημμένος. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Υπουργό και το προσωπικό του και θα υποδεχθούμε τον επόμενο Υπουργό. Allora prendiamo posto. Καθίστε παρακαλώ. Παρακαλώ όσοι θέλουν να παραμείνουν στην αίθουσα να καθίσουν. Να καλωσορίσουμε λοιπόν Καλημέρα σας λοιπόν. Ε, καλωσορίζουμε τον ε, Υπουργό Λεσόν, ο οποίος είναι Δανός Υπουργός ε, Επιχειρηματικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο μέχρι τη μία παρα Γι' αυτό λοιπόν στην ουσία μιλάμε για 42 λεπτά ακριβώς. Θα ήθελα να δώσω απευθεία το λόγο στον Υπουργό για την παρουσίασή του και κατόπιν θα συνεχίσουμε ο συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ σήμερα στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας αλλά θα ήθελα πρωτίστως ε, να συγχαρώ την Αμάλια Σαρτόρη για την ανάληψη των καθηκόντων της ως πρόεδρος της Επιτροπής και ε, προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία μαζί της. Από ό,τι βλέπω, πολλά από τα μέλη της Επιτροπής επέλεξαν να παραμείνουν μέλη της Επιτροπής και προσβλέπω λοιπόν και στη συνεργασία μαζί σας ε, στη διάρκεια της Ιτανικής Προεδρίας. Από πλευρά μα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας πάρα πολύ σημαντικό εταίρο. Έχουμε κοινέ εργασίε ε, οι οποίες μας περιμένουν και πραγματικά πρέπει να επιτύχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Η προτεραιότητά μας είναι ο συνεχής διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν και το έναυσμα για την ανάπτυξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Πολωνική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία επέτυχαν στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική συνεργασία μαζί τους. Η Δανία ανέλαβε τα ενία της Προεδρίας σε μια χρονική συγκυρία όπου βιώνουμε μια βαθιά κρίση και αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ. Ε, θέλουμε να αυξήσουμε την ε, δημοσιονομική και οικονομική συνεργασία και αυτό κυριαρχεί στο πρόγραμμά μας. Η Δανική Προεδρία λοιπόν θα προσπαθήσει να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους και ε, αντικειμενικούς σκοπούς που θα μας επιτρέπουν να έχουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία που χρειαζόμαστε για να έχουμε μια υπεύθυνη, δυναμική, πράσινη και ασφαλή Ευρώπη. Θεωρώ ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και η ανάπτυξη είναι οι δύο πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η Ευρώπη για να βγει από την κρίση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θα συνεργαζόμαστε για τους κοινούς μας στόχους και ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια Ευρώπη της ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ε, προχώρησε με τη Single Market Act που έχει βασικές πρωτοβουλίες τις οποίες θεωρούμε ότι θα συνεισφέρουν στην αύξηση της ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι περισσότερες από τις βασικές πρωτοβουλίες έχουν ήδη παρουσιαστεί και οι υπόλοιπες θα παρουσιαστούν στο εγγύς μέλλον. Η Single Market Act ε, θα συνεχιστεί στη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας και θα εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, χειροπιαστά αποτελέσματα στις περισσότερες από τις 12 βασικές πρωτοβουλίες και σε αυτό φυσικά θα έχουμε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Αυτές είναι η βασικότερη μεταρρύθμιση της ενίας αγοράς από το 1992. Και εγώ και η Ιδανική Προεδρία εν θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να υποστηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση. Πολλές από τις διατάξεις τη Single Market Art, κατ' εμέ συνεισφέρουν στον εξυγχρονισμό της ενίας αγοράς και συνεισφέρουν και σε μια πιο επικαιροποιημένη νομοθεσία, σύγχρονη, που θα μας επιτρέψει να έχουμε ως στόχο τον καταναλωτή, τον Ευρωπαίο πολίτη. Και μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο, ιδίω στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα και της ψηφιακής ενίας αγοράς. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τα σχέδια της Δανικής Προεδρίας για τον κανονισμό περιαγωγή 3, ε, ε, ε, την οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή και την οδηγία για την πρόσβαση σε δημόσια στοιχεία και επίσης θα ήθελα να σταθώ λίγο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο και την υπηρεσία ασφάλειας πληροφορικής, δηλαδή την ένισα. Η ψηφιακή ενέργορα είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται στην ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στους φραγμούς προς την ενέα αγορά και εξετάσαμε ευρύτατα το ζήτημα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να προάγουμε την ανάπτυξη ε, για τις ε, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Να μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρονικό εμπόριο διαμεθοριακά αλλά και για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν στο εξωτερικό με τα κινητά τους τηλέφωνα να μπορούν να έχουν κατάλληλες υπηρεσίες. Η δανική Προεδρία θεωρεί προτεραιότητα την ψηφιακή ατζέντα και θεωρούμε ότι αυτό είναι κοινό ενδιαφέρον και πολλών μελών εδώ της Επιτροπής σας. Πέραν αυτού, θα ήθελα να ζητήσω όσο το δυνατόν περισσότεροι από εσά να έρθουν στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου στην Κοπενχάγη 25 με 28 Φεβρουαρίου. Έχουν αποσταλεί προσκλήσεις προς τα μέλη της Επιτροπής και φιλοδοξία μας ε, είναι να προχωρήσουμε και τον κανονισμό για την περιαγωγή 3. Ελπίζουμε να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση στη διάρκεια της άναξης. Να υπάρχει δηλαδή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, διότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε επικοινωνίες μέσω κινητού τηλεφώνου είτε πρόκειται για ομιλία και σύντομα μηνύματα, SMS, όσο και για μεταφορά δεδομένων. Πρέπει να έχουν ευθυνή πρόσβαση σε όλες τις χώρες, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε να ρυθμίζουμε τα ανώτατα όρια των τιμών και ταυτόχρονα να ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα, ώστε ο ελεύθερος ανταγωνισμός να ε, λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Θα θέλαμε να επιτύχουμε ε, συμφωνία το συντομότερο το δυνατόν, και έχουμε και ε, διαπραγματεύσεις εν εξελίξη ε, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεργαζόμαστε μάλιστα και με την κυρία Νίμπνελ και με τους σκιώδεις εισηγητές επί του ζητήματος. Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ευθυγραμμίζεται με αυτό του Συμβουλίου. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό όταν ε, μας ενδιαφέρει το θέμα της ψηφιακής ατζέντα. Επίσης μας ενδιαφέρει το θέμα των υποδομών. Για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και πάλι στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε κατάλληλες υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πρόγραμμα για την, ε, το θέμα αυτό και συμπεριλαμβάνεται και στο Single Market Act. Ε, η πρόταση περιλαμβάνει ένα εγκάρσιο και φιλόδοξο νομοθετικό πακέτο. 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για προγράμματα επικοινωνίας ε, και για δημιουργία ψηφιακών υποδομών, για παράδειγμα πανευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών. Έγιναν οι αρχικές συζητήσεις στο Συμβούλιο και η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι χρειαζόμαστε πολύ στενό συντονισμό επί των ζητημάτων αυτών, διότι ε, οι διάφορες ομάδες του Συμβουλίου ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό ε, και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ισορροπημένα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μέσα τα οποία, τα κονδύλια συγγνώμη, τα οποία έχουν ανατεθεί θα χρησιμοποιούνται προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και της Ευρώπης εν γέννη και προς όφελος της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα τα οποία επιλέγονται για χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα προγράμματα ευρυζωνικών υποδομών, δεν θα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ούτε και σε επίπεδο κρατών μελών. Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πρόοδο και να διαπραγματευτούμε τα διάφορα στοιχεία της πρότασης ε, στον τομέα της πληροφορικής και της τηλεφωνίας. Ε, ε, συζητάμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές στην ομάδα του Συμβουλίου στην οποία προεδρεύω. Στο Single Market Act η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται και στις ηλεκτρονικές υπογραφές. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διαμεθοριακό και αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ενιαία αγορά και για τους καναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Και ελπίζουμε να έχουμε πρόταση από την Άνοιξη και να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από εκεί και πέρα να ε, παραδώσουμε τη σκητάλη στην Κυπριακή Προεδρία. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και η ε, σχετική οδηγία θα βελτιώσει το τοπίο για να υπάρχει πρόσβαση σε δημόσια αγαθά προς όφελος επιχειρήσεων είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματική νομοθεσία, διάφανη, να είναι πολύ καλά θεμελιωμένη από νομική σκοπιά και να μην υπάρχουν διακριώσεις ώστε να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός σε όλη την Ευρώπη. Έγιναν οι προκαταρκτικές συζητήσεις επί του ζητήματος αυτού στο Συμβούλιο και αναμένεται να είναι πολύ περίπλοκες οι συζητήσεις στο Συμβούλιο λόγω της εγκάρσιας φύσης της πρότασης. Μία από τις προκλήσεις είναι ότι ε, οι τροπολογίες που παρουσιάζονται αφορούν τους κανόνες ε, με τους οποίους καθορίζονται οι αμοιβέ για την περαιτέρω ε, εργασία δημοσίων δεδομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε περίοδο οικονομικής κρίσης να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Γι' αυτό και θα πρέπει να βρούμε μία ισοσχελισμένη λύση γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι δισταγμοί σχετικά με την ε, επέκταση του εύρους της ε, οδηγίας σε άλλα θέματα και θα προσπαθήσουμε να προβούμε σε αυτή τη διεύρυνση υπό την Δανεική ε, Προεδρία σε συνεργασία με τον εισηγητή κύριο Κάλφιν και τους Σκιώδης και διαπιστώνουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα διότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο λόγω της διαρκείας της εντολής και διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε χρόνο για να προχωρήσουμε. Ελπίζω ότι ε, η Δανική Προεδρία θα συμβάλλει και ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα συμφωνήσουν για να υπάρξουν εξελίξεις για το εγγύς μέλλον. Όπως ξέρετε ότι το Γαλιλαίο ε, είναι της αρμοδιότητος του Συμβουλίου Μεταφορών ε, και άρα ο συνάδελφός μου θα το χειριστεί αλλά του υποσχέθηκα ότι θα το αναφέρω εδώ σήμερα διότι το θέμα αυτό απασχολεί πολύ ε, τη ε, Ιδανική Προεδρία για την τεχνολογία της ε, πλοήγησης διαδορυφο... με τη βοήθεια δορυφόρων και θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την αυτιλία αλλά και για τις μεταφορές και η Δανική ε, Προεδρία έχει καθορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κατά τρόπον ώστε να επιτύχει μία μερική πολιτική συμφωνία πριν από το Συμβούλιο το αρμόδιο Συμβούλιο του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας, για την προθυμία σας να προβείτε σε διάφορες συμβιβαστικές λύσεις εν ώψη του ICT και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας είτε σήμερα είτε στο επόμενο εξάμεινο, όποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Έξι εγγεγραμμένους ομιλητές έχουμε και κατόπιν θα κλείσει ο κατάλογος. Μπένσεν, Thompson, Ρόμπικ Πουτικόφερ, Μπούζε και Βαλσίτης και κλείνει ο κατάλογος ώστε να δώσουμε και τρία λεπτά στον καθένα και έτσι θα μπορεί να απαντήσει και ο Υπουργός. Ο κύριος Μπένσεν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχά να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεδομένη τη τρέχουσα οικονομική κρίση είναι πάρα πολύ δύσκολο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει να λάβουν χρηματοδότηση για τι επενδύσει. Εσεί είπατε ότι πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και είπατε ότι το 80% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε προβλήματα γιατί ο τραπεζικός τομέας είναι και αυτός σε κρίση και είναι δύσκολο να υπάρξει χρηματοδότηση. Τον Δεκέμβριο η Επιτροπή δρομολόγησε ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήταν ένας από τους 12 πυλώνας, πυλώνες ε, της ε, ε, Παϊκής ενιαίας Πράξης και μήπως θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε πώς έχετε σκοπό να προχωρήσετε με το θέμα αυτό και πώς η πρόοδος πιστεύετε ότι θα γίνει κατά τη Δανική Προεδρία. κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Ε, προσβλέπω στο διάλογό μας ε, και με εσάς αλλά και με την Δανική Προεδρία στο σύνολό τη, ε, διότι η Επιτροπή μας καλύπτει πολλά θέματα. Μόλις κάποιος έκανε ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το θέμα αυτό είναι πολύ σχετικό με την ενιαία αγορά. Η 97% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού απασχολείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε προτεραιότητα στον τομέα αυτό τώρα. Όσον αφορά την ε, ενιαία αγορά, θα ήθελα να ρωτήσω για την, ε, για την ε, εξαγωγή των ε, υπηρεσιών έχουμε την ε, σχετική ε, οδηγία για τα προϊόντα, αλλά δεν έχουμε για τις υπηρεσίες. Και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε στην Ευρώπη εξάγοντας ο ένας τον άλλον. Υπήρξε και σεμινάριο σε σχέση με το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε την εξαγωγή των υπηρεσιών και πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό αν δεν κάνουμε τίποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα ζήτημα που, αφορά, που, που απασχολεί την ε, Δανική Προεδρία. Πολλές φορές έχουμε κάνει ε, αρκετά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την Δευτέρα, αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται πάντοτε γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα εργασιακό περιβάλλον ε, που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Υπήρξαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ε, με σκοπό την ενίσχυση ε, των συνθήκων ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να γίνουν και συνθήκες όμως φτωχότερες. Ευχαριστώ. Βέβαια εξελισσόμαστε σε ένα δανεικό μονοπόλιο όπως έγινε και στην ε, Ολομέλεια προχθές. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με ένα έγγραφο αξιολόγησης γιατί εγώ συνήθως είμαι στην αντιπολίτευση και δεν επενώ την κυβέρνηση αλλά πρέπει να πω ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία της Προεδρίας και έχετε συζητήσει και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις άρα η Δανική Προεδρία εκτιμά ιδιαίτερο στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο κατά τρόπον ώστε να έχουμε κάτι επιτυχές στο τέλος αυτής της πορείας της Προεδρίας. Ορισμένες προηγούμενες Προεδρίες υπήρξαν λιγότερο επιτυχής ακριβώς επειδή παραμέλησαν αυτή την πτυχή. Θέλω λοιπόν εδώ να αναφερθώ στο θέμα των διπλωμάτων ευρασίας ερασιτεχνίας και ε, μας ελέγχθη ότι βασίζεστε εις ε, τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά για να είμαστε ενιαία αγορά πρέπει να υπάρχει ενιαίο δίπλωμα ευρασιτεχνίας και θα πρέπει κάπου να μπορούμε να εντείνουμε τη συνεργασία. Η Ιδανική Προεδρία θα προσπαθήσει να προωθήσει το θέμα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι ένα στοιχείο με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ενία αγορά και θα προωθήσει και την εργασία στην Ευρώπη. Ο κύριος Μπιντικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ε, ε, σπάω τώρα το δανεικό μονοπόλιο και σας καλωσορίζω εξίσου θερμά στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω όμως ε, διότι η πολιτική μου οικογένεια συρίζει την κυβέρνησή σας αλλά όταν η αντιπολίτευση λέει ότι κάνετε καλή και έξυπνη εργασία δεν ξέρω τι μου μένει να πω εγώ αλλά εκτός από τα αστεία έχω να αναφέρω δύο θέματα σοβαρά. Το πρώτο αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά την περίοδο της προεδρίας σας θα χρειαστεί να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε διάφορα θέματα τα οποία είναι ε, αδύναμα σημεία, αδύναμη κρίκη και αναφέρονται στο ερευνητικό πρόγραμμα ε, της ε, Agenda του 2020. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο δεν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 ε, δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που θα έπρεπε να είναι η ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Βλέπουμε ότι 15% του προϋπολογισμού της ερεύνης πρέπει να καταλήγουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν έχει γίνει εφικτός ε, φιλόδοξος στόχος και βλέπουμε ότι στον προγραμματισμό για το 2020 μειώνεται και θα ισχύσει μόνο για τις προκλήσεις της κοινωνίας και τις τεχνολογίες και όχι όπου υπάρχει μία πραγματική αύξηση και άρα υπάρχει ο κίνδυνος οι επιχειρήσεις και ιδίω οι μικρομεσαίες με τη διεύρυνση αυτή του προγράμματος να μην ε, ε, λάβουν καμία χρηματοδότηση πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε τιμές του 2014 θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα χρήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι διατήθηκε ε, το 2007 σε τιμές του 2007 και ε, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό και θα πρέπει να το εξετάσει ένας υπουργός για την ανάπτυξη και να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την πορεία. Δεύτερον, στην Ευρώπη έχουμε μια ιδιομορφία της βιομηχανίας μας που σημαίνει ότι εξαρτόμαστε περισσότερο από τις αγωγές πρώτων υλών από ότι άλλα σημεία του ο κόσμου. Λέγεται ότι... Λέει ο ε, το Ποτοτσίν ότι 15 τόνους ανακεφαλήν ε, καταναλώνει ε, ο Ευρωπαίος πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν αυξηθούν οι τιμές οι τιμές για τον τελικό καταναλωτή θα επηρεαστούν πάρα πολύ και θέλω να ρωτήσω εάν πρόκειται να στηρίξετε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να εξευρεθεί μια κοινή λύση διότι ορισμένες χώρες έχουν ε, ε, ίδια προγράμματα και ε, εμποδίζουν, φρενάρουν και με τα δύο πόδια να προχωρήσει μια ενιαία πολιτική. Θα θέλα λοιπόν αυτή η ε, με συνεργασία να μπορέσει να προωθηθεί ιδιαίτερο υπό την Δανική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούζεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Υπουργό για τα εισαγωγικά, εισαγωγικά του σχόλια και για την παρουσία του. Θα ήθελα να συγχαρώ την Δανική Προεδρία για το πρόγραμμά της, ε, το πρόγραμμα Αναβίωση ε, της ευρωπαϊκής αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μας απασχολούν ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας ό,τι έχει να κάνει με τις ευρεσιτεχνίες, με την αναγνώριση των, ε, διπλωμάτων στο... στην ευρωπαϊκή αγορά, σημαίνει καλύτερη κινητικότητα για τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάρχει ένα μεγάλο κοινό πρόγραμμα και ο Επίτροπος Μπαρνιέ θέλει να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με την Δανική Προεδρία ε, θα είναι μεγάλη σημασία στην προσπάθεια αυτή. Το Κοινοβούλιο θέλει και εκείνο να συμμετέχει, γιατί η ιδέα της αναβίασης της ευρωπαϊκής ε, ενιαίας αγοράς προήλθε από το Κοινοβούλιο. Και ο κύριος Μόντι, ο Πρωθυπουργός της ε, Ιταλίας, ε, υπέβαλε τη σχετική πρόταση. Ο Δανός Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε θετικά και το ίδιο και ο Πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Παρόσο. Εξαρτάται όμως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα αποφασίσει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να εφαρμόζονται ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ταχαίω οι αποφάσεις. Έτσι είχε γίνει και στο παρελθόν. Ήταν πρόεδρο ο Ζακ Ντελόρ. πάλι κατόπιν ε, προτάσεως και πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια κοινή αγορά, μια κοινή αγορά ενέργειας είναι ε, βασικός παράγοντας. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή και με την Προεδρία. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω εσεί εκπροσωπείτε το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία που αφορά το δημοσιονομικό πακέτο και έχει να κάνει με την οικονομική διακυβέρνηση. Αφορά την οικονομία στην Ευρώπη. Ο τρόπο ε, ολοκλήρωση συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώ ε, σα κάνω τι εξή δύο ερωτήσει. Ιδανική Προεδρία έχει σκοπό να ε, συμπεριλάβει και χώρες εκτός ε, ε, Ευρωζώνης στις μελλοντικές συνόδους της Ευρωζώνης. Επίσης, εσείς ως Δανική Προεδρία θα επιτρέψετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως στις περχόμενες συνόδους. Εγώ πολλές εβδομάδες προσπαθώ να επιτύχω κάτι τέτοιο και νομίζω ότι θα ήταν κάτι το πολύ καλό για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μπαλτσίτης, τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς όρισατε κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστούμε πολύ για την πληρέστατη παρουσίαση του προγράμματος της Δανικής Προεδρίας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσά στο έργο σας, διότι το χαρτοφυλάκιο σας είναι πολύ περίπλοκο, περιλαμβάνει ε, σύγχρονες τεχνολογίες αλλά και πολλά άλλα θέματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση πρωτοβουλία. Στον 21ο αιώνα έχουμε χώρες, κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα εγκρίνει το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής και αυτό αποτελεί τεράστιο πρόσκομο για οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί όταν προτείνουμε συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική υπογραφή στις χώρες τους. Ένα ακόμα ερώτημα. Ο στόχος ε, διασύνδεσης της Ευρώπης ε, με διάφορα μέσα. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα και ορισμένες φορές δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλα τα προγράμματα ταυτόχρονα. Γνωρίζω από προσωπική πείρα ότι πολλές φορές γίνεται ανταλλαγή εγγράφων ε, μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών ή ακόμα και αυτοπροσώπως ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι αδιανόητο. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα στην ε, ε, στο Connecting Europe που θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ώστε να μην υπάρχει κατακαιρματισμός αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι παρεμβάσεις και οι ερωτήσεις. Ο λόγος τώρα για τα συμπεράσματα και τις τελικές απαντήσεις στον Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια και τα επικοδομητικά σχόλια, αλλά και τις ερωτήσεις. Καλά είναι τα πράγματα σε σχέση με τη συνεργασία μας ε, για τους επόμενους μήνες. Υπήρξε μία ερώτηση τον κύριο Μπένσον σε σχέση με τη χρηματοδότηση ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλοί θέσατε το θέμα της κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πώς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξή τους. Γιατί είναι ένα σημαντικό τομέα που επιφέρει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λοιπόν, η οδηγία για το κεφάλαιο κινδύνου είναι ιδιαίτερη προτεραιότητα στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας και θέλουμε να επιτύχουμε μία απόφαση σε πρώτη ανάγνωση στο πρώτο ήμιση του 2012. Και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει στο να καταλήξουμε συμφωνία γιατί αυτό θα είναι ιδιαίτερα υποφελέ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία που εγκρίνουμε υποστηρίζει το, στόχο μας ε, της ε, εξασφάλισης κεφαλαίου. Γι' αυτό ελπίζω να σημειωθεί πρόοδος προ αυτό. Υπήρξε επίσης μία ερώτηση για την οδηγία ε, για τις υπηρεσίες και για την εξαγωγή των υπηρεσιών. για τους ευφυείς κανονισμούς και πώς μπορούμε να επιτύχουμε ε, τα σωστά επίπεδα κοινωνικής προστασίας. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για ευφυείς ε, κανονισμούς. Πρέπει τα πράγματα να είναι όσο το δυνατόν σαφή και διαφανή και ε, πρέπει οι κοινωνικές συνθήκες ε, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών συνθήκων ε, δεν παραγνωρίζονται. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και αυτό μας απασχολεί ιδιαιτέρως και είναι βέβαια και πυρήνα της δουλειάς μας. Ο τρίτος συνάδελφος που πήρε το λόγο με τον οποίο σε εθνικό επίπεδο είχα πολύ καλές συζητήσεις Μιλήσατε για το θέμα των ε, τεχνιών. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε γιατί συμφωνούμε 100%. Είναι ουσιαστικό να λύσουμε το πρόβλημα της ευρεσιτεχνίας, ε, ο κανονισμός για τις ευρεσιτεχνίες ε, και είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει μεγάλο τμήμα της δουλειάς μας βέβαια συνεχίζοντας την τεράστια δουλειά της Πολωνικής Προεδρίας και τον ε, συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Εγώ επισκέφθηκα πολλές πρωτεύουσε, είχα πολλές διμερείς συζητήσει ε, στην αρχή της χρονιάς γιατί θέλουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι έχουμε τόσο κοντά φτάσει στο, στην ολοκλήρωσή του και γιατί τα ωφέλη μιας ε, κοινής, ενός κοινού συστήματος ευρεσιτεχνιών είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολλά. Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά στο τέρμα. Είναι δύσκολο ζήτημα, αλλά με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να πω ότι βασικοί παίκτες ε, υποσχέθηκαν ότι ενεργά θα συμμετέχουν για να μπορέσει να βρεθεί λύση στο, ε, κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Υπήρχε επίσης ένα ερώτημα σε σχέση με την φορολόγηση των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ο Υπουργός ε, Εσωτερικών ε, ασχολείται με τα θέματα αυτά, ή Υπουργός, και θα προτιμούσα να αφήσω την απάντηση σε εκείνη. Ούτως ή άλλως θα γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις και για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας. Υπήρχε και ένα ερώτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλοί έθεσαν το θέμα αυτό και το πρόγραμμα Horizon 2020 και το πρόγραμμα COSME έχουν έναν κοινό παρανομαστή κατά τη γνώμη μας και αυτό είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη. Το κόσμο είναι κάπως πιο ε, βραχυπρόθεσμο και προσπαθεί να βοηθήσει τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι πιο κοντά στην αγορά, ενώ το Horizon 2020 έχει ευρύτερη θεώρηση των πραγμάτων, την έρευνα, αφορά την έρευνα, την εκπαίδευση και είναι ένα πιο μακροπρόθεσμο εργαλείο ανάπτυξη. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε στα προγράμματα και στι προτεραιότητε αυτέ και ελπίζουμε ότι η Ιδανική Προεδρία θα μπορέσει να σημειώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στο πρόγραμμα ε, COSME. Πρέπει όμω να τονίσω ότι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών εξαρτάται στον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε επίσης ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, η σημασία της ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας έφερε στην οδηγία κεφαλαίου κινδύνου και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βασικές πρωτοβουλίες της οδηγίας για την ενιαία αγορά είναι και η βελτίωση της θέσει αλλά και των συνθήκων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, υπήρξε και ένα ερώτημα για το ε, οικονομικό πακέτο και ολόκληρη την κατάσταση γύρω από αυτό. Είναι ένα βασικό στοιχείο των διαπραγματεύσεών μας, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω περισσότερο για αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει προετοιμαστεί για την ανεπίσημη ε, σύνοδο τη Δευτέρα Και τέλος, για τις ηλεκτρονικές υπογραφές υπήρξε ένα ερώτημα. Βρήκα τις σημειώσεις μου γι' αυτό. Σε σχέση λοιπόν με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, θα ήθελα να πω ότι αυτό υπόκειται στο θέμα της ε, ψηφιακή ατζέντα και η Δανική Προεδρία θεωρεί ότι αυτό είναι τμήμα της προώθησης της ενιαίας αγοράς και γι' αυτό είναι και τμήμα των προτεραιοτήτων μας. Πιστεύουμε, είπαμε ότι θα ε, λάβουμε ανακοίνωση της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της Άνοιξης για το θέμα αυτό και ελπίζουμε να κινηθούμε με αυτό ως βάση και θα γίνουν και συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών ε, στις 8 ε, Ιουνίου. Σημειώνω επίσης τα σχόλια του κυρίου Μπαλτσίτης και θα ήθελα να του πω ότι έχουμε κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου επίσημο συμβούλιο για το θέμα αυτό και υπάρχει και στο τέλο του Φεβρουαρίου υψηλού επίπεδου διάσκεψη στην Κοπενχάγη για το θέμα αυτό. Είναι ένα εξαιρετική σημασία ζήτημα γιατί μπορούμε να δούμε δυναμικό ε, βελτίωση από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, ευχαριστούμε θερμά εξ ονόματο όλων των παρισταμένων, τον Υπουργό Σον και του συνεργάτε του για τη σημερινή του παρουσία εδώ και το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το εξάμεινο αυτό και για την Προεδρία να η Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά και τους διερμηνείς, διότι μας παραχώρησαν 10 λεπτά επιπλέον. Επόμενη συνεδρίαση, 6 Φεβρουαρίου, 3 με 6.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ εις το επανειδήν και ευχαριστούμε και πάλι τον Υπουργό και τους συνεργάτες του. Merci. À la prochaine Thank you. Hi. Hi.